Good morning, ladies and gentlemen. Please take your seats. Καλημέρα. Παρακαλώ, καθίστε για να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε με τις ψηφοφορίες. Μία ψηφοφορία έχουμε στρατηγική της Ένωσης για την περιοχή των Άλπαιων. Η συγητής είναι η κυρία Μπρέσο. Η συγητρία παρουσίασε την, ε, το σχέδιο συνεδρίασης στη συνεδρίαση του Απριλίου. Είχαμε λάβει 217 τροπολογίες. Επίσης, πρότεινε κάποιες συμβιβαστικές εσείς η κυρία. Θέλετε τον λόγο κυρία Μπρέσο πριν ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να πω δύο λόγια μόνο για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εργασία την οποία κάναμε. Συναντηθήκαμε πολλές φορές ε, ε, με τους σκιώδεις εισηγητές έτσι ώστε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις και νομίζω ότι ε, καταφέραμε να επιτύχουμε ένα κείμενο ευρεία συνενέσεως. Βεβαίως φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρξει κάποια διαφορετική ψήφος αλλά στο σύνολό τους νομίζω ότι οι κύριοι προβλήματα προβληματισμοί αντιμετωπίστηκαν και βρήκαμε επομένως κάποιες συμβιβαστικές λύσεις οι οποίες ε, επίσης ε, εμπλουτίζουν και το ίδιο το κείμενο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την, ε, το staff της Επιτροπής ε, γιατί ε, χρειάστηκε να εργαστεί πάρα πολύ. Ήταν πολλές οι τροπολογίες και επίσης αντίστοιχα πολλές και οι συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ωραία, να ψηφίσουμε λοιπόν. Και θα ξεκινήσουμε με την τροπολογία 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβασμός 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, απορρίπτεται. Τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 103 υπέρ κατά αποχές να εγκρίνουμε. Α, τροπολογία. Τροπολογία, έκανε λάθος η πρόεδρος. Τροπολογία ε, ε, 123. Τροπολογία 123. Ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Ζυχνόμη, λέει η πρόεδρος, έκανα λάθος. Πηγαίνουμε τώρα στο συμβιβασμό 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 127 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έχουμε εδώ μια προφορική τροπολογία, ωστόσο θα πάμε ε, στο συμβιβασμό 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται εγκρίνεται. Συμβιβασμός 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, ψηφίσαμε, ψηφίσαμε τη συμβιβαστική 30. 138 το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 144 υπέρ κατά 154 ε, εγκρίνεται. Έχουμε μια προφορική τροπολογία της εισηγητρίας. Ε, κάποιος αντιτίθεται σε αυτή την προφορική, όχι. Ψηφίσαμε λοιπόν με την προφορική τροπολογία. 155 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 159 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ. Α, υπάρχει ναι, ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 200 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 33, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 203, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 206, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 215 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 στις αιτιολογικές σκέψεις, ε, αναφορές, συγγνώμη, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5, για την αιτιολογική σκέψη α. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6, αιτιολογική σκέψη β. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 36, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, σκέψη σκέψεως Β, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 επί της ιδεολογικής σκέψεως C υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Εδώ έχουμε προφορική τροπολογία. Κάποιος αντιτίθεται στην προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν τη 16 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ καλά, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 επί της αιτιολικής σκέψεως C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ είναι προφορική τροπολογία. Κάποιος αντιτίθεται, όχι, επομένως ψηφίζουμε την τροπολογία 23 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 25 ε, για την ιδιωτική σκέψη ή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 επί της αιτιολογικής σκέψεως F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πηγαίνουμε τώρα στις ε, προτάσεις της ε, ε, Επιτροπής Απασχόλησης, ΕΜΠΛΑ A. Κυρία Μπρέσο, θέλετε να πείτε κάτι. Να σας πω ότι εγκρίναμε πολλές από τις προτάσεις των Επιτροπών ε, ήδη στις συμβιβαστικές τροπολογίες ε, και αυτό ίσως εξηγεί κάποιες αρνητικές ψήφους. Επαναλαμβάνω πολλά από τα στοιχεία που είχαν προτείνει οι Επιτροπές τα έχουμε ήδη ενστερνιστεί. Ήταν σημαντική πραγματικά, σημαντικό πραγματικά να, πούμε γιατί ε, απορρίψηθηκαν κάποια πράγματα. Εκτός μικροφώνου παρατηρήσει οι διερμηνείς δεν ακούν. Εξακολουθούν να μην ακούν οι διερμηνείς, παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου δυστυχώς. Πρόεδρος, εντάξει, θα προσπαθήσω να, τα, να κάνουμε τις ψηφοφορίες από κοινού, unblock. από το A μέχρι το K υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται ε, L Α, είναι συμβιβαστική. Ωραία, καταπίπτει λόγω της συμβιβαστικής. Προτάσεις M, η M, η L είπαμε καταπίπτει. M, N, O. Ναι, αλλά θα πρέπει για τα πρακτικά να, να πούμε τι κάνουμε. Από το M μέχρι το 18 ψηφίζουμε λοιπόν εκτός από αυτά που καταπίπτουν υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Προτάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κλπ. Με τον ίδιο τρόπο θα ψηφίσουμε από το A μέχρι το C en μπλοκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβιβασμός 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε από την πρόταση E μέχρι τη συμβιβαστική 35 εκτός αυτών που καταπίπτουν υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι προτάσεις από την 25 μέχρι την 32 υπέρ κατά αποχές και αυτές απορρίπτονται. Προτάσεις τώρα από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού μπορούμε να κάνουμε το ίδιο, δηλαδή να ψηφίσουμε από την πρόταση A μέχρι την πρόταση 14 πλην όσων καταπίπτουν υπέρ παρατηρήσεις εκτός μικροφώνου. Ε, στις άλλες φορές δεν υπήρχε πρόβλημα, αλλά τώρα... C suggestion. Is that correct? Ε, A to C is fine. Από το A μέχρι το C μπορούμε. Ε, ε, λοιπόν, ε, η πρόταση A υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πρόταση B υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και πρόταση C υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται Απορρίπτεται. Τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε on block. Εντάξει, αλλά θα πρέπει να μου λέτε ποιες είναι αυτές που θέλετε να ψηφίσουμε χωριστά. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Συμβιβασμός, ε, συγγνώμη, πρόταση D. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Πρόταση E. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, πολύ ωραία. Πρόταση D, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ποιαν θέλετε να επαληθεύσουμε, την D, την D, ωραία, D, D όπως ο Δούναβης, Δέλτα. Πέρας της ψηφοφορίας. και απορρίπτεται. Σε πρόταση Ή e, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. F υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. GH 1, 2, 3, 4 καταπίπτουν. Να ψηφίσουμε από κοινού 5 μέχρι 13. Ωραία, 5 μέχρι 13, εκτός από αυτές που καταπίπτουν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Και τώρα έχουμε τις προτάσεις Επιτροπής Γεωργίας. Θα κάνουμε χωριστή ψηφοφορία ή unblock. Μέχρι την 24 Μέχρι την 24 λοιπόν μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού. Όχι. Πρόταση παριθμών 1 καταπίπτει λόγω της... Λοιπόν, συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 5 καταπίπτει. 6 υπέρ κατά αποχές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 απορρίπτεται. Η 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 24 καταπίπτει, η 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 29 καταπίπτει 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας Συγχαρητήρια κυρία Μπρέσο. Αν κρίνεται η έκθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay, ladies and gentlemen, we can... Ωραία, ναι, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Το επόμενο θέμα είναι ανταλλαγή απόψεων για τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 όλα τα τμήματα. Και χαίρομαι που καλωσορίζω εδώ πέρα σήμερα τον κύριο Γιάνς Γκάιερ, τον Γενικό Εισηγητή για τον Προπολογισμό του 2017. Ο κύριος Γκάιερ θέλει να συνεργαστούμε για τους, ε, πολιτικ... για τους φακέλους πολιτικής συνοχής γύρω στο 1 τρίτο του συνόλου Γι' αυτό είμαστε στις ε, συζητήσει Σήμερα λοιπόν θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και μια παρουσίαση του σχεδίου, του σχεδίου περιπολισμού των Κομισιόν που όπως ξέρετε έχει αναπληθεί από το τέλος Μαΐου για το τέλος Ιουνίου. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Βόν, δεν είναι εδώ πέρα σήμερα και ο κύριος Νίλσεν θα παρουσιάσει την γνωμοδότησή του, αλλά λίγο αργότερα όχι τώρα. Τώρα θα δώσω λόγο στον κύριο Γκάιερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε σήμερα το πρωί για τον προϋπολογισμό για το έτος 2017. Έχω την τιμή να προετοιμάζω την πρόταση του προπολισμού εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος φέτος θα τα κάνουμε κάπως διαφορετικά από ό,τι συνήθως γιατί το είπατε η Κομισιόν ανέβαλε την δημοσιοποίηση του προϋπολογισμού κατά τέσσερις εβδομάδες. Κατά κανόνα ήταν στο τέλος Μαΐου η Κομισιόν είπε ότι χρειάζεται ακόμα χρόνο για τον επανυπολογισμό των δαπανών για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Βεβαίω το ότι η προθεσμία αυτή είναι μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα προφανώς δεν έχει ούτε μία σχέση, αλλά ο Γενικός Διευθυντής ο αρμόδιος το επιβεβαίωσε αυτό και την Δευτέρα, ότι δεν έχει ούτε μία σχέση με το Βρετανικό δημοψήφισμα. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν πλέον προσέχει και να μην χτυπάει τις πόρτες δυνατά πως τρομάξουν οι Άγγλοι. Και Κάτι παρόμοιο είχαμε και το 2014 πριν τις ευρωεκλογέ, μια αναβολή. Οπότε το θέμα του πόσο γρήγορα θα σχηματίσει και θα καταλήξει μια θέση στο Συμβούλιο είναι πλέον το ανοιχτό ζήτημα. Και αυτό οδήγησε στο ότι χθε αποφασίσαμε στην Επιτροπή Υπερπολογισμού να γίνει ο πρώτος διάλογος ε, αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτά είναι τα οργανωτικά προβλήματα. Βεβαίως έχουμε και τα χρηματικά. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές ε, που αποφασίσαμε στην Ολομέλεια του Απριλίου τα που καθορίζουν τα επιχειρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χοντρικά και ξεκινήσαμε με αφετηρία και είδαμε πως ε, υπήρχε μεγάλη στήριξη το ότι οι ανάγκες του 2017 δεν θα είναι πολύ διαφορετικές από αυτές του 2016 και κυρίως έχουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετα που κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση και όσον αφορά τις αιτίε, αλλά και για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την εισρωή. Αυτό σημαίνει πως οι κατηγορίες 3 και 4 για εσωτερική και εξωτερική πολιτική, δηλαδή αντιστοίχως, εξαντλήθηκαν μέχρι το πλαφόν που επέτρεπε ο κανονισμός και δεν βλέπω εγώ κάποια αφορμή να που με κάνει να πιστεύω ότι θα έχουμε μείωση των αναγκών το 2017. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα αποθεματικά μας στις δύο αυτές κατηγορίες πλέον δεν υπάρχουν και δεύτερον, επειδή οι κατηγορίες του προπολογισμού ε, σχεδόν δεν ε, καλύπτονται με μια τεχνική εξαίρεση που είναι πολύ περίπλοκη, δεν μπορούμε να διαθέσουμε ε, κονδύλια από άλλες κατηγορίες για τις 3 ε, και 4. Θα είναι μεγάλη η συζήτηση με το Συμβούλιο γιατί βεβαίως πάντα η προσπάθειά τους είναι να κινηθούν, να αφήσουν ένα περιθώριο μεταξύ του πλαφών το πολιετού προγράμματο και των ετσίων ε, προπολογισμών, γιατί λένε ότι πρέπει να έχουμε κάποιο απόθεμα, αλλά και για να μην ε, εγκρίνουν πολύ ψηλέ πληρωμέ εκ των προτέρων. Ένα πρόβλημα το οποίο θα έχουμε στον προπολογισμό αυτόν είναι πως όλες ε, οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που του παρελθόντος εξακολουθούν να ισχύουν και έχουμε και την ε, χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων που είναι και 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο έτος 2017 και στα επόμενα βεβαίως. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το ποσό για το Ταμείο Γιούνκερ το λεγόμενο κάπως θα πρέπει να βρεθούν λοιπόν αυτά τα δισεκατομμύρια. Όλα αυτά δείχνουν κατά την άποψή μου πως το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο όπως είχαμε αποφασίσει το 2013 ήταν αυτό το οποίο λέμε ότι θα λειτουργούσε υπό κάπα σίγμα, αν τα πράγματα δηλαδή πήγαιναν χω... χωρίς προβλήματα. Αλλά με τις ε, συνθήκες αυτές ένα τεράστιο κύμα προσφύγων ε, το μεγαλύτερο από τον δεύτερο παγκόσμιο, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οπότε... Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την συζήτηση στο νέο, για το νέο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίση, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Κομισιόν να συνδέσει τον Προπολογισμό στενότερα με τα μέσα τα οικονομικά που έχει η Κομισιόν στην διάθεσή της. Έχουμε λοιπόν τις τελευταίες οικονομικές προοπτικές, την έκθεση για την ανάπτυξη, την διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτά τα μέσα λοιπόν της Κομισιόν θα πρέπει να αξιολογηθούν. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μια δημοκρατική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά να αποφασίσουμε ποια από αυτά τα οποία μας προτείνει η Κομισιόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε στον προπολογισμό επιπλέον. Πρέπει να δούμε και τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Ε, θα ήθελα να αναφέρω δύο από αυτούς που με απασχολούν εμένα ιδιαίτερα. Το ένα είναι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων με τη σχετική πρωτοβουλία και, ε, άλλο ένα βεβαίως ε, και αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα περιβάλλον πολιτικό δύσκολο, αυτό το οποίο γνωρίζετε και μια κατάσταση στο Συμβούλιο όπου δεν έχουν και πολύ όρεξη να διαθέσουν λεφτά, αλλά στην πορεία θα διαπιστώσουν ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό είναι το πλαίσιο θα έλεγα και αναμένω τα δικά σας τα σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τις ε, εισαγωγικές παρατηρήσεις σας για να ξεκινήσει η συζήτηση. Νίλσεν τώρα παρακαλώ για να παρουσιάσει τη θέση του κυρίου Βόν που είναι εισηγητής μας στην Επιτροπή Ρέγγι. Έχετε τον λόγο. Ελπίζω ότι είναι στην Ουαλία, στην εκστρατεία για την παραμονή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια σημεία μου ε, κατέγραψε και θα σας τα αναγνώσω με τη δική του διατύπωση. Ίσως σχολίαζε ο ίδιος τα όσα είπε ο Γκάια. Αλλά αυτά έχουμε και που είναι σημαντικά ενώπιόν μας τώρα για την Επιτροπή Ρέγγιο η σημασία της ε, δράσης ε, της ε, Επιτροπής μας ως Επιτροπής η Επιτροπή Συνοχής αποτελεί την κύρια επένδυση στην πραγματική οικονομία για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή. Γι' αυτό ο προπολογισμό του 2017 είναι πολύ σημαντική υπόθεση και πρέπει πολύ προσεκτικά να εξεταστεί. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν επαρκή κονδύλια στον προπολογισμό, ιδιαίτερα στην κατηγορία 1β, για να αντιμετωπιστούν όλες οι υποχρεώσει πληρωμών σε σχέση με τα διαδοτικά ταμεία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των μη επαρκών πληρωμών που δημιουργεί προβλήματα. Ο προπολογισμό 2017 πρέπει να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε ένα σωστό πρόγραμμα και σχέδιο. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σημειώσει πρόοδο στην απλούστευση των κονδυλίων, των διαδικασιών διάθεση των κονδυλίων, ιδιαίτερα για να ανακουφιστεί η επιβάρυνση των υποφελούμενων, των εμπλεκόμενων σε αυτά τα σχέδια. Πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα στις δράσεις μας να βρούμε τρόπους να μετρήσουμε την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων ώστε να αξιολογήσουμε πού δαπανήθηκαν καλά τα χρήματα και πού δεν δαπανήθηκαν σωστά και πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις. Είναι σημαντικό να είμαστε αποτελεσματικοί για εξοικονομήσεις ώστε να χρησιμοποιούμε κάθε ευρώ αποτελεσματικά. Δίνοντας μάχη για το μέλλον της πολιτικής συνοχής πρέπει να δείξουμε ότι είναι αποτελεσματική και κάνει τη διαφορά. Επίσης σημειώνουμε ότι περισσότερα κονδύλια πιθανότητα, πιθανότατα θα πρέπει να διασφαλιστούν για τους ε, μετανάστες και πρόσφυγες. Και έτσι αυτό μέσα στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020 και του μηχανισμού διασύνδεσης της Ευρώπης που πρέπει η χρηματοδότησή τους ε, να φτάσει στα παλαιότερα επίπεδα. Είναι σημαντικό να, για την παρουσίαση της Επιτροπής στην 27η Ιουνίου, αλλά στις 13 Ιουλίου 2016 θα έχουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και έτσι θα μπορέσουμε να καταθέσουμε τις τροπολογίες μας μέχρι την 20 Ιουλίου 2016 αν χρειαστεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σκιώδης εισηγητές για παρέμβαση, για τη γνωμοδότηση, όσοι επιθυμούν να παρέμβουν. Δεν βλέπω την κυρία και Ο κύριος Φανίστερ Ρόι, εξ ονόματος του ΕΛΚ, παρακαλώ. Υποστηρίζω την προπαρασκευή που έγινε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για αυτό το θέμα. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις σε αυτό με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και τον εισηγητή Κάθε χρόνο ουσιαστικά επαναλαμβάνεται αυτή η διαδικασία. Το Συμβούλιο τίνει να αποκαταστήσει εκείνα που χρειάζονται για την περιφερειακή πολιτική όσο αφορά τον προϋπολογισμό, εκείνα τα κονδύλια που χρειαζόμαστε. Μπορούμε να βασιστούμε λοιπόν σε αυτή την παλαιά οσήθιστε μέθοδο που ακολουθούμε για να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι επενδύσεις στην Επιτροπή Συνοχής στα επίπεδα που είχαμε συμφωνήσει παλαιότερα. Και αυτό είναι το κυριότερο βέβαια. Δεύτερο επίσης, όσον αφορά τις νέες εξελίξεις, νεότερες εξελίξεις, ε, όπως το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε ότι έχει καλές επιδόσεις στο Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Στρατηγικών Επενδύσεων και θα μπορούσε να επεκταθεί, να παραταθεί. Αυτό που θα θέλαμε είναι πιο εξειδικευμένα με στοιχεία κατά λεπτό στα αποτελέσματα αυτού του νέου μέσου του ΕΤΣΕ. Υπάρχουν ε, κάποια πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά τους πολλαπλασιαστές. Ε, είναι απίστευτο αυτό που λένε ότι υπάρχει 16 απλάσιος λέει πολλαπλασιαστής ή πάνω και από 20, 20, 20 Δεν μπορούσα ποτέ να κατανοήσω πώς μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Γενικά τετραπλάσιος ο πολλαπλασιαστής, ένα ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για παράδειγμα, αποκινούμε επενδύσεις ε, από το εθνικό επίπεδο, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και οι ιδιώτες επενδυτές μπορεί να καταλήξει σε 4 ευρώ, τετραπλάσιο αποτέλεσμα. Αλλά όλοι λένε εντάξει, ωραία, αν υπάρχουν κονδύλια, δάνεια έστω, ε, τότε μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά εγώ γνωρίζω ότι το δάνειο πρέπει να επιστραφεί, να αποπληρωθεί. Καλό είναι να υπάρχει η ροή ε, κονδυλίων, αλλά σε τέτοιες συγκυρίες ε, είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε τα πράγματα. Γι' αυτό η Ευρωκοινοβουλευτική μας Επιτροπή θα πρέπει να εργαστεί εξετάζοντας βαθύτερα τα μέσα και τους τύπους των μέσων τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν υπάρχει αποτυχία της οικονομίας ή της αγοράς σε πάρα πολλά πράγματα δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές ώστε να υπάρξει ανάπτυξη στην έρευνα για παράδειγμα και να υπάρξει για παράδειγμα στις περιοχές σύγκλησης αντίστοιχη δράση. Δεύτερο, είναι υπέροχο βέβαια ότι 100 δις ας το πω έτσι, ρευστοποιούνται όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων και διατίθενται. Είναι σαν την πρόγνωση όμως τη μετεωρολογική. Μπορεί να βρέξει εδώ ή αλλού την επαύριο, την ε, επόμενη μέρα. Ε, μπορεί να συμβεί το ένα ή το άλλο. Δεν υπάρχουν κάποια τεκμήρια, αποδείξεις πίσω από τέτοιες υποθέσεις ε, σε σχέση με μια θεματολογική προσέγγιση. Πώς θα γίνουν όλα αυτά. Δεν είναι ακριβώς επακριβή λοιπόν σε σχέση με τον προπολογισμό 2017. Θέλω να κάνω αυτή την προειδοποίηση. Χρειαζόμαστε τεκμήρια για αυτά τα κύρια επενδυτικά ρεύματα, τα κύρια επενδυτικά μέτωπα και επιπρόσθετα να δούμε επιπρόσθετα μέσα τα οποία δημιουργούνται τώρα και πώς λειτουργούν και ποια αποτελέσματα έχουν. Αυτά θα ήθελα να υπογραμμίσω. Ότι χρειαζόμαστε σίγουρα καλές ε, τεκμηριωμένες εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προβληματιστούμε σε βάθος για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και εμείς με βάση όλα αυτά. Εφόσον λοιπόν είναι ασαφή τα πράγματα και είναι ασαφή για μένα όσον αφορά θέματα της Επιτροπής Ανάπτυξης πρέπει να βασιστούμε στο πλαίσιο του προπολογισμού έχει για την περιφερειακή πολιτική. Είναι αναγκαία αυτά τα κονδύλια, τα χρειαζόμαστε τα επόμενα χρόνια πρέπει να διατεθούν. Τα λειτουργικά προγράμματα τα οποία βρίσκονται υπό εξέλιξη, υπό δρομολόγηση, πρέπει να μπορέσουν να προχωρήσουν. Καθυστερήσαμε πραγματικά ξεκινώντας αυτά τα νέα προγράμματα. Όμως τα καλά μαντάτα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε σε σχέση με τα 25 δις που θα μπορούσε να διαθέσει σε ένα ας το πω έτσι αποδεκτό επίπεδο το αποτέλεσμα είναι εκείνο που πρέπει να δούμε σε σχέση με τα κονδύλια για τη νέα περίοδο. Και προβλέπω ότι θα υπάρξει μια εντονότατη ροή κονδυλίων ε, μη εξοφλούμενων ε, λογαριασμών του χρόνου και θα επαναληφθεί αυτό και το 2018 και 2019 φοβούμε. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά ικανοποιημένοι λοιπόν και ευτυχεί για μια τέτοια κατάσταση. Λέει η Επιτροπή πετύχαμε το στόχο. Ναι, στρεφόμενοι προ τα πίσω. Είναι σημαντικό να εξοφλούνται οι λογαριασμοί, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση για το μέλλον. Ίσως και το αντίθετο μπορεί να υπάρξει και θα υπάρξει ενδεχόμενα πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Σα ευχαριστώ που ήρθατε εδώ για να καλυφθεί το έργο αυτό όπω πρέπει. Ευχαριστώ. Κυρία, Κυρία είσαστε σκιώδη εισηγήτρια. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. The right balance between fiscal consolidation. Όλα αυτά που μας είπατε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Στηρίζουμε ε, λοιπόν έναν ε, λογικό προϋπολογισμό για το 2017 που θα ισορροπεί ανάμεσα ε, στην δημοσιονομική πρόνοια αφενός και τις σωστές επενδύσεις αφετέρου. Βεβαίως χρειάζεται σωστή αξιολόγηση των αναγκών που θα πρέπει να βασιστεί σε καλές δημοσιονομικές πληροφορίες. Επίσης ε, πρέπει να υπογραμμιστεί ή ε, ε, να υπογραμμιστεί η ανάγκη τροποποιητικοί προϋπολογισμοί να παραμείνουν στο ελάχιστο έτσι ώστε έγκαιρα τα κράτη-μέλη να μπορούν να υπολογίσουν τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι ο επόμενος σκιώδης εισηγητής. Θα πάρω λοιπόν το λόγο εξ της ομάδας μου Άλντε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Γκάιερ για την ανταλλαγή ε, απόψεων που γίνεται σε ένα πολύ πρόημο στάδιο και χωρίς να έχουμε και την πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να έχουμε ε, την ε, γενική κατεύθυνση του Κοινοβουλίου για την Άλντε, για την πολιτική μου ομάδα. Είναι ε, σημαντικό στον προϋπολογισμό του 2017 να δούμε συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία είναι διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και τα, ε, ε, και τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής αλλά και το Ταμείο Επενδύσεων ΕΦΣΥ. θα πρέπει ο σχεδιασμός να είναι καλός, η διεύθυνση να είναι ε, καλή και ο προϋπολογισμός να ε, έχει στόχο την αποτελεσματικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεύτερον, αναφέραμε ότι δουλεύουμε ε, για τον προϋπολογισμό 2017 ταυτόχρονα με την εργασία μας για την αναθεώρηση των πολιετών ε, ε, προοπτικών. Δουλεύουμε επομένως ταυτόχρονα για τον προϋπολογισμό του έτους αλλά και για το πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε τις κύριες κατευθύνσεις της μεταρρύθμισης και της αλλαγής του πλαισίου και να δούμε αυτές τις αλλαγές να υλοποιούνται στον προϋπολογισμό 2017, γιατί αυτός θα είναι ο προϋπολογισμός ο οποίος θα υπογραμμίζει, θα παρουσιάζει ε, όλα τα νέα ζητήματα, τους νέους προβληματισμούς που δεν, ε, είχαν, που δεν ε, υπήρχαν στον ορίζοντα όταν προετοιμάσαμε το προηγούμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Θα πρέπει να αποφευχθούν ε, οι δημιουργίες προβλημάτων και αδιεξόδων τα επόμενα χρόνια. Ε, είναι γεγονός επίσης ότι έχουμε ε, μικρά κεφάλαια χρηματοδοτήσεων όσον αφορά τα επιχειρησιακά προγράμματα. Επομένως όλα αυτά τα μέτρα τα οποία θα μας βοηθήσουν να αποφύγουμε αδιέξοδα ή ε, προβλήματα τα επόμενα χρόνια ε, είναι κάτι θετικό και θα πρέπει να αντικατοπτριστούν οπωσδήποτε στον προϋπολογισμό του 2017 δηλαδή ήδη να περιληφθούν και στον προπολογισμό και στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Επίσης, θέλω να υπογραμμίσω ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα βρίσκονται ακόμα ε, σε αρχική φάση υλοποίησης, αλλά το 2017 αναμένουμε τα πραγματικά αποτελέσματα, τις πραγματικές επιπτώσεις των νέων πολιτικών και των νέων επιχειρησιακών ε, προγραμμάτων. Και αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη του ο προϋπολογισμός του 2017. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ και μίλησα εξ ονόματος της ομάδος Άλντε. Ο κύριος Ομάρ Ζε είναι ο επόμενος ε, ε, σκιώδης, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Ομάρ Ζε. Είμαστε συνάδελφοι στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και είμαι μάλιστα και σκιώδης εισηγητής επί της ε, ε μεταρρυθμίσεως του πολιετούς ε, χρηματοδοτικού πλαισίου. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ο προϋπολογισμός και το πλαίσιο είναι δύο θέματα τα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν εκ παραλίλου. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι για να επιτύχουμε τους στόχους μας θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε σωστές ισορροπίες δυνάμεων σήμερα με το Συμβούλιο ε, και αυτό θα έχει επίπτωση οπωσδήποτε και στο ρυθμό προώθησης ε, των αποφάσεων για τον προϋπολογισμό 2017. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και για όλους είναι ότι επιλέξαμε να μην περιμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αναφέρουμε και να επιβεβαιώσουμε τους δικούς μας ε, προσανατολισμούς και όσον αφορά την αναθεώρηση του πλαισίου και για τον προϋπολογισμό του 2017. Το Κοινοβούλιο λοιπόν λέει ότι είναι δύο έγγραφα τα οποία έχουν μεγάλη πολιτική δύναμη με την έννοια ότι ε, καταδεικνύουν πρώτο, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχα την ευκαιρία να το ξαναπώ, αλλά το βλέπουμε κάθε χρόνο πόσο αυτός ο πολιτικός πολιετής ε, προϋπολογισμός είναι δεσμευτικός και το 16 και το 17 μιλάμε για προϋπολογισμούς που στην ουσία ε, δεν επιτρέπουν ή οριακά ε, να απαντηθούν τα ερωτήματα ή τα ζητήματα τα οποία έχουν ε, παρουσιαστεί. Έχουμε εξαντλήσει κάθε όριο αποθεματικού και κάθε όριο ευελιξίας για το 2016 και δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Αυτό φαίνεται και στις συζητήσεις και φάνηκε και στις συζητήσεις που είχαμε για τον προϋπολογισμό που θεωρούσαμε ότι είναι ε, ε, προϋπολογισμός λιτότητας που δεν είχε σαφώς την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Το είχαμε πει από πριν, το κατανοούμε πλέον σαφώς και νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους όταν θα ξεκινήσει ή μάλλον όταν θα τοποθετηθούν στη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του πολιετούς πλαισίου. Όσον αφορά το προϋπολογισμό, το θέμα των πληρωμών είναι κάτι σημαντικό για το 2017, θα γίνει ακόμα πιο βαρύ για το 2018, γιατί οι πραγματικές ε, πληρωμές ε, τότε θα ξεκινήσουν και θα πρέπει ο προπολογισμό να είναι προετοιμασμένο. Υπάρχει και κάτι που δεν αφορά μέσα τον προπολογισμό 2017, αλλά θα πρέπει να πάρει θέση η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και αναφέρομαι στην διάρκεια του προπολογισμού. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις ε, έτσι ώστε ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεω να είναι πενταετής και όχι επταετής. Ε, που ταυτίζεται με τη διάρκεια των προγραμμάτων. Έχει ξεκινήσει ε, μια μεγάλη συζήτηση και θα ήθελα ο εισηγητής να μου πει την άποψή του επί του θέματος αυτού. Να σας πω ότι εγώ προσωπικά έχω κάποιες ανησυχίες Εάν δηλαδή ε, ε, με προβληματίζει λίγο το να μειώσουμε ε, την διάρκεια και να μην ταυτίζεται με τη διάρκεια του πλαισίου, γιατί φοβούμε ότι έτσι θα προσθεθούν επιπλέον δυσκολίες στις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες συνοχής όσον αφορά ας πούμε την ΚΑΠΑ. Το 2017 εν ολίγης, για μία ακόμα φορά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ στενό, πολύ σφιχτό προϋπολογισμό με μία κατάσταση η οποία ε, μέρα με τη μέρα αποκαλύπτει τα προβλήματά της, αποκαλύπτεται ως πιο δύσκολη Επίσης έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις στην ε, Επιτροπή μας όσον αφορά την Ελλάδα έτσι ώστε να τις επιτρέψουμε να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες και αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει, για την Ελλάδα θα πρέπει να ε, ε, συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό. Κύριος Λόπε. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα τα σχόλιά μας να σας αναφέρω για τον προϋπολογισμό του 2017. Φυσικά κάθε φορά όταν συζητούμε θέματα προϋπολογισμού βλέπουμε ότι οι απαιτήσει στα αιτήματα είναι υψηλότερα από τις δυνατότητες και όταν έχουμε κρίσεις υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση κονδυλίων. Και όταν σχεδιάζουμε τον προϋπολογισμό είναι τεράστια σημασία να έχουμε τις σωστές προτεραιότητες και είναι πολύ σημαντικό στη συνέχεια να χρηματοδοτηθούν αυτές οι προτεραιότητες επαρκώς. Δεν επαρκεί να υπάρχουν απλώς προτεραιότητες που θα έχουμε διατυπώσει. Είναι σημαντικό να χρηματοδοτηθούν όπως πρέπει αυτές οι προτεραιότητες. Και είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό των 5 δις ευρώ για το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη έχουν τώρα τη δυνατότητα αυτή και μπορούν να την ακολουθήσουν. Όμως θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτό το ταμείο θα πρέπει να εργαστεί ώστε να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, οι διαφορές που υφίστανται σήμερα. Διότι τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ότι χρησιμοποιείται μόνο από κάποια κράτη-μέλη το ταμείο αυτό. Και μάλιστα έχουν πολύ μεγάλα προγράμματα και σχέδια που χρηματοδοτούν από αυτά τα κονδύλια αυτού του, του ταμείου μεγάλους αυτοκινητοδρόμους ε, και αυτό δεν θα δώσει κοινωνική συνοχή, απλώς θα αυξήσει τις υποδομές ε, για τις μεταφορές και τις διασυνδέσεις της πόλης μας. Η ενεργειακή αποδοτικότητα, η ενεργειακή απόδοση, η, η χρήση των ορυκτών ε, καυσίμων, και η υποκατάσταση τους θα πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτείται από το Ταμείο αυτό και να υπάρχουν και γεωγραφικά κριτήρια και στόχοι για το Ταμείο. Να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου μόνο μόνο ή 10 κράτη-μέλη θα απορροφούν και έτσι θα εξαντλούν τα κονδύλια αυτού του Ταμείου και δεν θα απομένει τίποτα για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειαζόμαστε κάποια όρια, κάποια ανόφλια. Πρέπει να θέσουμε τέτοια περιθώρια ώστε να, επιτρέπονται, να επιτρέπεται σε περισσότερα κράτη-μέλη να κάνουν χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και να διασφαλίσουμε επίσης ε, να, ότι θα μειωθούν οι διαφορές μεταξύ περιφερειών στα κράτη-μέλη. Ένα άλλο θέμα τώρα, το θέμα των προσφύγων. Φυσικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει. Όμως φυσικά αυτό απαιτεί κονδύλια πάλι που πρέπει να εξευρεθούν. Πρέπει να καθορίσουμε τα αναγκαία ποσά που πρέπει να διατεθούν. Και επιπρόσθετα σε όλα αυτά, εγώ ως πρώην δήμαρχος, που γνωρίζω και μπορώ να σας πω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να ενταχθούν οι νεοαφιχθέντες, οι επίλυδες ε, σε μια πόλη. Αυτό δημιουργεί πιέσεις και προβλήματα. Πρέπει να διασφαλιστούν λοιπόν κονδύλια για αυτό το στόχο, για τις περιφέρειες. Οι περιφέρειες θα πρέπει να κάνουν προσαρμογές στα προγράμματά τους και στα κοινωνικά προγράμματά τους προγράμματα επίσης για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια τα οποία είναι αναγκαία για την ένταξη των προσφύγων ε, στο κοινωνικό περίγυρο, στην κοινωνία. Όλα αυτά κοστίζουν πολλά. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ και ελπίζω να ληφθεί αυτό υπόψη. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο, τον κύριο Σιλίβ να πάρει το λόγο, καθώς επίσης και τον κύριο Λέιβ Οβρες. Ποιος θα πάρει το λόγο? Παρακαλώ. Φίλιπ Ζωέ, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω σε σχέση με αυτά που εξήγησε ήδη ο Γενικός Εισηγήτης. Βεβαίως η Κομισιόν δεν έχει φτάσει ακόμα στο τελικό ε, σχέδιο προϋπολογισμό που όπως είπατε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος γιατί θα πρέπει να συμφιλιώσει, να συντονίσει, να συνδυάσει διάφορα προβλήματα, διάφορες κρίσεις. Ε, προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε με το μέγιστο βαθμό ευελιξία, αλλά παρόλα αυτά, ε, που, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει στα πλαίσια του MFF, του πολιετούς χρηματοδοτικού ε, πλαισίου. Ε, αυτά τα ανέφεραν άλλωστε και οι διάφοροι ομιλητές. Είναι γεγονός ότι όσον αφορά τον τομέα των ε, πληρωμών ε, είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε ξεπεράσει το ε, πρόβλημα με τις πληρωμές που δεν έχουν ακόμα καταβληθεί. Βεβαίως θα πρέπει να προσέξουμε το 2017, να προσέξουμε όλα τα στοιχεία για τις, για τις πληρωμές ε, σε σχέση με όλα αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως. Όλα τα προσέχουμε, ε, αλλά προσέχουμε βεβαίως ε, και το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα τα οποία θα συμπέσουν με το τέλος του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Κύριε Γκάγερ, θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου σε κάποια από τα θέματα που προαναφέρθηκαν να τοποθετηθώ. Καταρχήν η κρίση πληρωμών. Εγώ είμαι στην ευτυχή θέση να μπορώ να πω ότι στον επόμενο προϋπορισμό αυτό δεν θα μας πλήξει ιδιαίτερα. Δεν θα μας αφορά ιδιαίτερα. Κάποιοι συνάδελφοι το προανέφεραν. Είναι ένα πρόβλημα που κατά το τέλος της περίοδου πληρωμών μπορεί να παρουσιαστεί πάλι το εξηγώ αυτό έτσι, ότι έχουμε τραβήξει την κουβέρτα μέχρι το λαιμό μας. Έχουμε αποφύγει τον κίνδυνο να κρυολογήσουμε, όμως κρυώνουμε, τα πόδια μας κρυώνουν επειδή έχουμε τραβήξει την κουβέρτα ψηλά. Αυτό σε σχέση με την, ε, τις, ε, τα προβλήματα το 18, 19, 20 ίσως υπάρξει κάποια τέτοια κατάσταση. Είμαι πιο αισιόδοξο ότι μπορούμε όμως να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτή την κατάσταση διότι προς μεγάλη μου έκπληξη δίωσα διαπραγματεύσεις ε, πληρωμών του προϋπολογισμού όπου το Συμβούλιο αριθμητικά μεγέθη ποσά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα αμφισβητούσε. Είχε υποβάλει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν ε, θα δεχόταν. Με αυτή τη βάση φυσικά πολύ δύσκολα μπορούν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις. Αυτό το έχουμε αποφύγει, το αποφεύγουμε τώρα. Επειδή σε τακτά διαστήματα έχουμε τριμερείς διαλόγους και επανεξετάζονται τα ποσά αυτά αμέσως. Αν δούμε λοιπόν ότι πληρωμές ε, και αποθεματικά δεν επαρκούν, τότε το Συμβούλιο, νομίζω το προπροηγούμενο έτος ε, το έμαθε το Συμβούλιο αυτό, όταν έπρεπε να δώσει πρόσθετα 3,3 δις με άλλα λόγια, πιστεύω ότι τώρα σε σχέση με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου υπάρχει περισσότερος ρεαλισμός πλέον σήμερα για αυτά τα θέματα. Αλλά να πω το εξή η πολιτική του Συμβουλίου επί μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό αντανακλάται μεσοπρόθεσμα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να μην δουν μόνο τις υποχρεώσεις, αλλά να βλέπουν τις πληρωμές που βρίσκονται απέναντι στις υποχρεώσεις. Στις υποχρεώσεις δεν έχουν προβλήματα, ακολούθησαν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Όμως κλείνουν το πουγγί όταν έρθει η ώρα των πληρωμών. Δεν τα διαθέτουν. Και θεωρητικά σε σχέση με την Επιτροπή Περιφερικής Ανάπτυξης, συζητώντας με τους πραγματογνώμονες, κάθε πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιαστεί δεν μπορεί έτσι να υλοποιηθεί. Κάποια αποβιώνουν, αποθνίσκουν καθοδόν σε σχέση με τα μεγάλα προγράμματα υποδομών που ε, δεν πρέπει να καθυστερήσουν, έλεγε το Συμβούλιο, αλλά δεν χρειάζονται αυτά τα κονδύλια ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως δεν μπορούν σε αυτό το πλαίσιο να υλοποιηθούν σε αυτές τις διαστάσεις. Μπορώ να φανταστώ 1%, 0,5% των πληρωμών σε σχέση με τις υποχρεώσεις να παραμείνει. Εντάξει, αλλά 4-5% συστηματικά περικοπές δεν γίνεται και έχουμε αυτή τη διάθρωση σε σχέση με τα πολιετή δημοσιονομικά προγράμματα διότι έχουμε δεσμεύσεις για 950-960 δις ευρώ που όμως υποχρεώσεις 907 δις βρίσκονται απέναντι. Έχουμε διαφορά 50 περίπου δις. Και αν στην περιφερειακή πολιτική, και αυτό είναι, αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες ε, σε σχέση με τις δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που πρέπει να είναι πολιτικός μας στόχος, δηλαδή να μπορέσουν το δυνατόν τα περισσότερα προγράμματα να υλοποιηθούν, είναι σαφές ότι με μια τέτοια κατάσταση, με μείωση, με απουσία 50 δισεκατομμυρίων, δημιουργούνται πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχουμε τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης τώρα και μπορούμε αντίστοιχα να δράσουμε για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, αλλά ο κίνδυνος να καταλήξουμε σε μια τέτοια κρίση δεν έχει αποκλειστεί τελείως Έχουμε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης όπως είπα, αλλά οι πληρωμές όσον αφορά υποχρεώσεις ε, πληρωμών και την εκτέλεσή τους ε, είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται. Και δεν πρόκειται μόνο για κονδύλια και ποσά στον όγκο τους, αλλά και για την ποιότητά τους. Πρέπει να αναβαθμίζεται αυτή. Η Επιτροπή συζητά έντονα το θέμα των επιδόσεων στον προϋπολογισμό performance based budget. Έχει νόημα αυτό. Δεν έχει νόημα απλά να έχουμε κάποια χρήματα για να γίνει μια γέφυρα κάπου, όλα να πηγαίνουν και να βαίνουν καλώς, να γίνονται οι προκηρύξεις, να μην υπάρχει κάποιο σφάλμα, ποσοστό σφάλματος, αλλά η γέφυρα να χτίζεται σε λάθος τοποθεσία ή να μην μπορεί έτσι να χρησιμοποιηθεί. Στην, επιτρο... στην ε, δημοσιονομική συζήτηση αυτό δεν είναι χωρίς σημασία η ΕΠΑ για παράδειγμα ε, πολύ λίγο ελέγχει το ελεκτικό συνέδριο εκεί τη συμμόρφωση compliance βλέπει το θέμα της, ε, των επιδόσεων performance ε, και σε σχέση με τα ποσοστά σφάλματος που γίνεται μεγάλη συζήτηση πάντα σε σχέση με εμά, όλα αυτά αποσύρονται για να διεξάγεται μια ποιοτική συζήτηση. Τι πετυχαίνουμε με τα κονδύλια του προϋπολογισμού και ποια είναι η ποιότητα αυτών που επιτυγχάνουμε, αυτό πρέπει να δούμε. Και ακριβώς ε, δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη δική μας ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πρέπει να βοηθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι σωστές συνιστώσεις και παράμετροι ώστε στα πολυάριθμα προγράμματα και σχέδια που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης να μπορούμε να μετρήσουμε το βαθμό και ποσοστό επιτυχίας. Αν προβληματιστούμε επ' αυτού, ε, συνάδελφοι, είναι σαφές ότι στις επιδόσεις, performance, θα ασκήσει μοχλευτική πίεση το Συμβούλιο και θα πει υπάρχουν αυτές οι αναβαθμίσεις ε, διότι διαφορετικά να κάνουμε ε, ε, τέτοια προγράμματα τα οποία θα έχουν αναβαθμισμένη ποιότητα. Θα είναι λοιπόν φλέγον αυτό το θέμα και όσο νωρίτερα προσαρμοστούμε σε αυτή την πραγματικότητα τόσο το καλύτερο. Επόμενο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι το θέμα του ΕΦΣΥ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Ναι, ο Κατάινεν την τελευταία φορά μας το πέρασε, μας το πούλησε ως επιτυχία. Ερώτημα είναι όμως αυτά δεν θα ήταν προγράμματα και σχέδια που θα χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ούτως ή άλλως. Δεν απαντήθηκε όμως αυτό το ερώτημα από πλευράς του. Και φυσικά συζητώντας με τους επαΐοντες, τους πραγματογνώμονες, η εγγύηση για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν αυτά που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν για την περιφερειακή ανάπτυξη είναι κάτι σημαντικό. Θα πετύχουμε αυτό το οποίο επιθυμούμε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, δηλαδή σορευτικότητα δεν φαίνεται να το πετυχαίνουμε κάτι τέτοιο με την κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Και αναφέρθηκε από τον συνάδελφο Ρουπέ και αφορά και τη Γερμανία σχετικά. Φυσικά ωραίο είναι αν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων χρηματοδοτηθεί, χρηματοδοτεί αυτοκινητοδρόμου στην Γερμανία. Αλλά ο Υπουργό Οικονομικών λέει ωραία τέλεια δεν έχουμε ελλείμματα, έχουμε σημείο ε, που έχουμε εξισορροπήσει έσοδα δαπάνε. Ε, πρέπει σε σχέση με την λεπτή διαχείριση των, των κονδυλίων να έχουμε και την αρχή της ε, αθρηστικότητας ή σωρευτικότητας και να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά καλύτερα. Εγώ είμαι υπέρ των διαβουλεύσεων ώστε η ποιότητα των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σχεδίων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στατικών Επενδύσεων να βελτιωθεί. Μια επικοδομητική συζήτηση για το ΕΤΣΕ αξίζει να διεξαχθεί λοιπόν υπό αυτούς τους όρους. Και σκέφτομαι διαζώσεις τώρα, εκφράζοντας τις σκέψεις μου με αυτά που σας λέω. Αν για παράδειγμα χρήματα που στις εγγυήσει θα μπορούσαν από το έτσι να εγγραφούν, εμείς αν δεν θα έπρεπε αυτά να τα θέσουμε στο αποθεματικό μέχρι ότου να μεριμνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξουν κάποια πράγματα από πλευράς του ΕΤΣΕ. Δηλαδή θα εγγράψουμε κονδύλια, αλλά θα μπουν στο αποθεματικό, θα τροχοπέδι, θα παγώσουν δηλαδή και θα απελευθερωθούν μόνο όταν θα έχουν υπάρξει τα αποτελέσματα εκείνα που θα έχουμε ζητήσει εμείς. Και θα δούμε υπό ποιους όρους στο μέλλον θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεύτερο, και α, τούτο θέλω να πω ως ε, αρμόδιος για τα δημοσιονομικά, για την κρίση προσφύγων. Έχω πικραθεί κάπως για την κατάσταση που όπως έχει διαμορφωθεί τι κάνει το Συμβούλιο. Υπό οποιοδήποτε σχηματισμό το Συμβούλιο έχει φιλόδοξες δεσμεύσεις που κάνει, ποια χρηματοδοτικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιηθούν, ποια κονδύλια, ώστε με το Ταμείο για την Αφρική, για, με, την, το μέσο, με την Τουρκία για τους πρόσφυγες, ώστε το πικρό πεπρωμένο των προσφύγων να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και να βοηθήσουμε. Έρχεται μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει «Α, εδώ υπάρχουν μεγάλες ε, δεσμεύσεις. Κάποια μετάθεση πρέπει να γίνει στον προϋπολογισμό ώστε να διασφαλιστούν οι πληρωμές». Και το έκανε και το Συμβούλιο και αυτό. Και βλέπω τι ροέ κονδυλίων σε σχέση με τα κράτη και αγαπητοί συνάδελφοι, πραγματικά είναι σχρή κατάσταση. Απαράδεκτη κατάσταση. Γίνονται μεγάλε υποσχέσει από τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ω δημοσιονομική αρχή, παράλληλα με το Συμβούλιο, κάνουν τη δουλειά του όταν πρόκειται για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη που πρέπει να προσθέσουν από πλευρά του κονδύλια για να συμπληρώσουν αυτά τα κονδύλια για την διευκόλυνση για την Τουρκία πρόκειται για μια αναλογία 2 προ 1 δεν κάνουν τίποτα. Με 3 εκατομμύρια εντάσσονται στο Ταμείο το ελάχιστο ποσό που θα διασφαλίζει ότι θα μπορεί να υπάρξει δυνατότητα ε, μετάθεσης ή ε, αποσυμφόρησης και μετά δεν κάνουν τίποτα. Δεν δεν είναι το θέμα λοιπόν της δέσμευσης κονδυλίων καθοδών ε, εν ρευστό. Πρέπει να δούμε τι είναι πρόθυμα να πληρώσουν τα κράτη-μέλη και εμείς να πληρώνουμε τα άλλα 50%. Δεν θα δεχθώ περισσότερο να δίνουμε 250 εκατομμύρια εμείς στον προϋπολογισμό για την πρώτη δόση της διευκόλυνσης για την Τουρκία και από τα κράτη-μέλη με κάποια διψήφια ποσά εκατομμυρίων να παίζουν το παιχνιδάκι τους. Ναι, χρειαζόμαστε τα χρήματα διότι δεν είναι η ροή ε, ε, στην ε, πρώτη φάση αρκετά ισχυρή αλλά αν αυτό ισχύει και ισχύει για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πρέπει να δούμε τι πληρώνουν τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να πληρώνουν τα υπαρκή κονδύλια. Και όταν θα το κάνουν, τότε θα ακολουθούμε και εμείς από πλευρά μας με τις αναγκαίες πληρωμές από τη δική μας πλευρά. Αυτά θέλω να πω και κυρία Τούμασιτς, σε σχέση με την ε, ε, κοινοβουλευτική ομάδα δεν θέλω να εξαιρέσω κάποιον από τα όσα λέω. Αν το Συμβούλιο δεχόταν να γίνουν αυτά θα το βλέπαμε αλλά το αίτημά σας τότε μόνο μπορεί να υλοποιηθεί αν το Συμβούλιο της ΕΕ <clears throat> δεν παραμένουν καθοδόν διαρκώς ε, παρουσιάζοντας νέες ιδέες πώς πρέπει να γίνει το ένα ή το άλλο και αλλάζοντας τους όρους του παιχνιδιού. Τι θέλω να πω. Θα ήμουν ευγνώμων πραγματικά αν μπορούσαμε να αντιμετωπίζαμε τα πράγματα όπως πρέπει. Μόνο που δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε προβλέποντας τις κρίσεις, όλες τις κρίσεις παγκόσμια. Και ως υπεύθυνο για τα χρηματοοικονομικά, τα δημοσιονομικά, αντιμετωπίζω την κατάσταση ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αντίδραση στην κρίση, τι έχουμε, χρησιμοποιούν κονδύλια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες. Και μετά σκέφτονται τι θα μπορούσαν οι ίδιοι τα κράτη-μέλη να κάνουν για να αντιμετωπιστεί συμπληρωματικά η κατάσταση ρεαλιστικότητα και προβλεψιμότητα για ένα σχεδιασμό που θα ήταν αναγκαίος με αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να τεθούν αυτοί οι όροι στο Συμβούλιο και να πούμε να διοποιηθούν αυτά ώστε να, να επομίζεται το Ευρωκοινοβούλιο τις ευθύνε του. Αλλά πρέπει να κάνει τη δική του δουλειά το Συμβούλιο. Δεν μπορεί να αφήνεται μια κατάσταση με κάποιες αναλύσεις να συντάσσουν μια συνταγή πώς θα προχωρήσουν παραπέρα αλλά να στέλνουν το λογαριασμό που πρέπει να πληρωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να λένε ότι εμείς ε, που, εμείς που έχουμε τόσα πολλά χρήματα πρέπει εμείς να υπομισθούμε αυτές τις ανάγκες, τις πληρωμές. Αν σταματούσε το Συμβούλιο με αυτή την πρακτική τότε θα πετυχαίναμε αυτό το οποίο απαιτού, απαιτείται, δηλαδή προβλεψιμότητα σχεδιασμού. Και θα ήμουν ικανοποιημένο αν θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί. Εφόσον όμως συνεχίζεται αυτή η πολιτική, φοβούμαι ότι θα, είμαστε, θα παραμείνουμε απογοητευμένοι. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκατε ακριβώς στον προϋπολογισμό με βάση την απόδοση και τη σχετική συζήτηση, η δική μας η Επιτροπή και έχουμε πολλές εκθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ακριβώς κάνει. Στον νέο κανονισμό έχουμε ακριβώς ε, αυτή την θεματική εστίαση, όχι δηλαδή γέφυρες στο πουθενά, στα πράγματα αυτά που θέλουμε να εργαστούμε, γνώση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνικά, υπολογιστές τηλεπικοινωνίε και μέσα στα προγράμματα μετά έχουμε τους δείκτες αυτούς ε, της απόδοσης. Έτσι δουλεύουμε τώρα. Και κάναμε μάλιστα και ένα αποθεματικό απόδοσης 6% των χρημάτων μας που θα δοθεί σε αυτούς που τα πάνε καλά. Οπότε έχουμε αλλάξει ε, ουσιαστικά. Δηλαδή αν υπάρχει καμία γέφυρα στο πουθενά είναι από το παρελθόν, από παλιά προγράμματα. Τώρα στη νέα αυτή περίοδο που χρησιμοποιούμε την μέθοδο αυτή νομίζω πως Έχουμε ένα καλό παράδειγμα και για άλλου ε, τομείς πολιτικής, όπω η αναπτυξιακή πολιτική που δεν δουλεύει καθόλου έτσι. Ε, μπορούμε να αποδείξουμε στα επόμενα έτη, 16-17 ειδικά, αλλά και τώρα, στην έκθεση την 16.3, ότι έχουμε αποτελέσματα. Οπότε υπάρχει μια καλή βάση για μια κοινή συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κλείνει εδώ η συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Είμαστε στη διάθεσή σας με την γνωμοδότηση του κυρίου Βόνη και για περαιτέρω συνεργασία. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Συνεχίζουμε τώρα με την μερίσια διάταξη. Το επόμενο θέμα είναι η γνωμοδότηση κυρίου Πορέμπα και αφορά την νομοθετική έκθεση της ε, Επιτροπής Βιομηχανίας για έναν κανονισμό που αφορά μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο. Η Επιτροπή μας αποφάσισε να συντάξει μια γνωμοδότηση. Οι άλλες επιτροπές είναι η ΑΦΕΤ, η ΕΚΟΝ, η ΕΜΚΟ και η ΤΡΕΝ. Ο εισηγητής μας τώρα θα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης και προτείνω οι τροπολογίες να κατατεθούν μέχρι της 22 Ιουνίου. Τον λόγο έχει ο κύριος Πορέμπα για να παρουσιάσει την έκθεσή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την πολύ σημαντική αυτή γνώμοδότηση. από την ε, έγκριση του κανονισμού το 2010 όταν σημειώθηκε κάποια πρόοδος για την ολοκλήρωση των αγορών αερίου που μας επέτρεψε να εισαχθούν κάποια μέτρα ασφαλείας. Νομίζω πως ε, η εμπειρία μας μέχρι σήμερα δείχνει Ειδικά αν σκεφτούμε τις ε, κρίσεις του 2006, του 2009 και του 2014, όλες αυτές οι εμπειρίες μας δείχνουν πως μιλάμε για διασυνοριακά ζητήματα που επηρεάζουν ολόκληρη την Ένωση και οι κανονισμοί αυτοί ελάχιστα προστατεύουν τις εγχώριες αγορές και με τρόπο πολύ περιορισμένο. Και με τεχνικούς όρους Νομίζω πως ε, αντιμετωπίζουμε γενικότερα προβλήματα περιφερειακής ε, υφής και πολιτικά επίσης. Και νομίζω πως, και θέλω να το τονίσω αυτό, πως ε, είναι πάρα πολύ θετικό το ότι η προτεραιότητά μας είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Και αυτός είναι ένας στόχος ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό μιλάμε ακριβώς για την ασφάλεια εφοδιασμού και για το ότι θέλουμε ακριβώς να έχουμε αυτά τα μέσα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Και βεβαίω είμαστε υπέρ ε, των προτάσεων που εστιάζουν στην αρχή της ε, αλληλεγγύης, ε, την διαχείριση κινδύνου και προσπαθούμε βεβαίω να ξεπεράσουμε αυτούς τους κινδύνους. Επίσης κάποιες περιφερειακές ομάδες μας δείχνουν το τι μπορεί να γίνει για να βελτιώσουμε την ασφάλεια εφοδιασμού και έτσι θα γίνει ο κανονισμός ε, πιο αποτελεσματικός. 90% των ε, ροών αερίου στην Ευρώπη είναι διασυνοριακές και αυτό σημαίνει πως Υπάρχει κίνδυνος οποιαδήποτε αναταραχή να μεταδοθεί. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται πολύ στενή συνεργασία και συντονισμός. Θεωρώ πως η περιφερειακή αυτή προσέγγιση που προωθώ και στηρίζω εγώ είναι επίσης ε, πάρα πολύ ε, σημαντική και βεβαίως ε, Υπάρχει και το ζήτημα των συνεπειών της κρίσης ε, στην Ένωση. Τα διαφανή κριτήρια και συγκεκριμένοι μηχανισμοί συνεργασίας οπωσδήποτε θα οδηγήσουν σε μια διαφοροποίηση των πηγών το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία σε περιπτώσεις ανάγκης και νομίζω πως ε, ο καλύτερος περιφερειακός ε, συντονισμός, ο οποίος βασίζεται σε κοινέ προδιαγραφές που θα εγκριθούν στο επίπεδο της Ένωσης, δίνουν στα κράτη-μέλη πραγματικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τους ε, κινδύνους ε, που σχετίζονται με την υπερβολικά υψηλή ζήτηση ή την χαμηλή παροχή. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός για να παρέχεται αέριο στα νοικοκυριά ε, και στα νοσοκομεία παραδείγματο χάρη και σε άλλους οι οποίοι παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες. Εις βάρος προφανώς άλλων πελατών. Και βεβαίως θα τονίσω στην εκθεσή μου το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών και θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ειδοποιείται αυτομάτως ε, για σημαντικές συμβάσεις αμέσως μετά την υπόγραφή τους και οι αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αιτιολογημένα να ζητούν πληροφορίες για να αξιολογούν τους κινδύνους ε, εφοδιασμού για να υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια. Αναμένω λοιπόν την γνωμοδότηση αυτή και ελπίζω να έχουμε μια γνωμοδότηση η οποία θα αναφερθεί στους μηχανισμούς ε, για το πώς θα διασφαλίσουμε επαρκές αέριο για τα κράτη-μέλη ειδικά σε περιπτώσεις ανάγκης. Αυτός θα πρέπει να είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους μας, να φροντίσουμε δηλαδή η περιφερειακή διάσταση να διατηρηθεί και να την στηρίξει η Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο, στους ο κύριος Αχμαν είναι εδώ, ο κύριος Βανίστερο, εξ του ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Χάκμαν δεν είναι εδώ. Αλλά πολύ με την παιδική σας προσέγγιση. Να κάνω μια πρώτη παρατήρηση. Το φυσικό αέριο Ε, είναι θεμελιώδες στοιχείο της, ε, του ενεργειακού ε, μείγματος. και στη μετάβαση την οποία προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε το φυσικό αέριο, το οποίο είναι φυσικά πολύ καλύτερο από το άνθρακα. Και νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια θα εξακολουθεί να είναι σημαντικό το φυσικό αέριο. εξαρτάται πολύ, όπως το λέτε και εσείς, η Ευρώπη από τις ε, εισαγωγές αερίου. Ο νέος κανονισμός, ε, λοιπόν, είναι εξαιρετικά σημαντικός και ε, καταδεικνύει και τα ασθενή σημεία όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού. Το 2006 ας πούμε, το 2009, το 2014 ήταν χρόνια κρίσης όσον αφορά τον εφοδιασμό ε, και δεν θα είναι και τα τελευταία. Όπως είπατε, η δημιουργία περιφερειών είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό θέμα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να γνωμοδοτήσουμε και εμεί ως Επιτροπή. Ε, η περιφερειοποίηση βεβαίως εδώ ε, είναι πολύ μεγαλύτερο, μεγαλύτερης κλίμακας, όχι απλά ενεργασία μεταξύ δύο περιφερειών. Επίσης ο κ. Χάρτμαν θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι ε, χρειάζεται αλληλεγγύη με τους γείτονες ε, για να αντιμετωπιστούν έκτακτες καταστάσεις. Και σε αυτό το σημείο τα μαθήματα είναι πολλά. Μπορούν να γίνουν πολύ εύκολες αλλαγές. Πριν από δέκα χρόνια ε, τα οι βενζινοπόλες στα βενζινάδικα μπορούσαν να έχουν μόνο ε, μονή ροή, μονής κατεύθυνσης ε, μέχρι πριν από 10 χρόνια. Η δυνατότητα αντίστροφης ροής λοιπόν μπορεί να ακούγεται απλό αλλά είναι μεγάλη σημασία. Δεύτερον, υποχρεώθηκαν τα κράτη-μέλη να έχουν στρατηγικά αποθέματα γιατί σε περίοδο κρίσης, ας πούμε, ή έλλειψης, ε, τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει το κράτος τη δυνατότητα να αντλήσει από κάποια επιπλέον ε, αποθέματα. Επίσης, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ε, διαφάνεια. Διαφάνεια, λοιπόν, όσον αφορά τα μέτρα. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Αλλά ε, μετά από πόσο διάστημα, μετά από ποια ημέρα προβλήματος ε, οφείλεις να στηρίξει τον γειτονά σου. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν. Επίσης, ο κύριος Χάρτμαν... Συμφωνεί με τις τροπολογίες σας, ε, μάλλον με τη γενική σας προσέγγιση, αλλά ε, θα υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την θέση που παίρνει το ΕΛΚ για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μόρκοβα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε... Σας ευχαριστώ. Θέλω την, να αφήσω εκτός την πολιτική παρουσίαση η ανάλυση οι προλαλήσαντες εξήγησαν γιατί είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η ασφάλεια τροφοδότησης ε, εκ νέου. Κάποια μαθήματα ε, μάθαμε από το παρελθόν, τα όσα αναφέρθηκαν από πλευρά του συμφωνώ με τις παρατηρήσεις σε τρία πράγματα που είναι σημαντικά πρέπει να επικεντρωθούμε. Πρώτον, και προαναφέρθηκε αυτό, στην περιφερειακή διασύνδεση θα πρέπει από αυτήν να εκινήσουμε. Οι χώρες που βρίσκονται σε διαφορετικές περιφέρειες χρειάζονται καλές σχέσεις μεταξύ τους. Πρέπει να έχουν καλά ανεπτυγμένες υποδομές και ταυτόχρονα κάθε περιφέρεια θα πρέπει με το σωστό ισορροπημένο τρόπο θα πρέπει να ε, συμμετέχει σε σχέση με το κράτος της ε, η περιφερειοποίηση δεν μπορεί να είναι ένα εμπόδιο στη διμερή συνεργασία μεταξύ κρατών η σύνθεση των περιφερειών είναι σημαντική υπόθεση. Τα κράτη-μέλη στόχευαν στο να υπάρξουν κοινά προγράμματα και σχέδια και πρέπει οι υποδομές εφόσον υφίστανται να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο, να υπάρξει ένα εναρμονισμός, να υπάρξει μια διασύνθεση διαδρόμων. Επόμενη παρατήρηση, ο μηχανισμός αλληλεγγύης και αυτό αναφέρθηκε προηγούμενα. Έχω την εντύπωση ότι είναι αναγκαίο να αποσαφινιστούν τα πράγματα επακριβώς, ώστε να είναι σαφές ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εταίρων όσον αφορά την αλληλεγγύη μεταξύ τους, όταν υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν είναι αποκλειστική υπόθεση των κρατών αυτή. Πρέπει και η Επιτροπή να τοποθετηθεί σε σχέση με τις υποχρεώσεις υπονομικό πλαίσιο όσον αφορά αυτές τις συναλλαγές, αυτό το εμπόριο. Επόμενη παρατήρηση σε σχέση με το άρθρο 5 για τη συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου. Θα πρέπει να υπάρξουν επακριβέστερες διατυπώσεις και προτάσεις. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει να αποσαφινιστεί πλήρως να αποκλειστούν κίνδυνοι, ενδεχόμενα κινδύνων. Η γειτονία προς την Ουκρανία σε σχέση με την αγορά φυσικού αερίου ο όγκος του φυσικού αερίου είναι πολύ μεγάλος. Ε, δεν είναι το ίδιο με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες γειτονικές χώρες, για παράδειγμα, γειτονικές χώρες της Ουκρανίας. Στην Ανατολική Ευρώπη πρέπει τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται όταν υπάρχει διακοπή παροχής φυσικού αερίου. Και ο νέος ορισμός ε, των ε, θεμελιωδών κοινωνικών υπηρεσιών. Και εκεί βλέπω να υφίστανται κάποιες δυσκολίες. Διότι θα πρέπει να, υπάρξει να υπάρχουν προστατευμένες ομάδες ευάλωτες ομάδες που θα προστατεύονται. Υπάρχουν όμως και επιφυλάξεις ε, κρατών μελών ε, για τέτοια θέματα. Είμαστε πρόθυμοι σε σχέση με τις, την κατάθεση τροπολογιών να προχωρήσουμε με αυτή τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για τον σκιώδη εισηγητή κύριο Γιάκο η παροχή φυσικού αερίου αποτελεί τμήμα της συνολικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ενεργειακά θέματα που θα προωθεί την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το 2010 έγινε ένα πρώτο βήμα για ένα διευρυμένο συντονισμό ώστε να αντιμετωπίσουμε την διασυνοριακή πρόκληση της ε, ε, διασφάλισης παροχής ε, φυσικού αερίου. Υπάρχουν όμως οι διαφορές ε, των κρατών μελών και ο διασυνοριακός χαρακτήρας και πρέπει να άρουμε τα εμπόδια μεταξύ κρατών μελών αλλά επίσης να έχουμε χαμηλότερο κόστος πρόληψης. Σε σχέση με την περιφερειακή λοιπόν προσέγγιση από πλευρά των κρατών μελών που ήδη σχολίασε αυτό το θέμα ο κύριος Φανίστερ Ρόι σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση από πλευρά μας αυτή η περιφερειακή προσέγγιση για τα ενεργειακά θέματα και την ενεργειακή ασφάλεια είναι πολύ σημαντική υπόθεση για την, ε, τον επιμερισμό ε, του φυσικού αερίου ανάλογα με τις ανάγκες μας διευρύνοντας ε, την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανθεκτική, απαιτεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της παροχής φυσικού αερίου από εγγενείς πηγές Χρειαζόμαστε τη βελτίωση της αποδοτικότητας και πολυμορφοποίηση όσον αφορά την εξάρτησή μας από εξωτερικές πηγές. Και η Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να στοχεύουν σε αυτήν την πολυμορφοποίηση όσον αφορά την ενεργειακή μας τροφοδότηση και την παροχή αυτών των αγαθών. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με θέματα ενεργειακής ασφάλειας και από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και από πλευρά κατών μελών. Προγράμματα που δεν ανταποκρίνονται σε αυτέ τι προδιαγραφέ δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατευθυντήριε γραμμέ δεν πρέπει να είναι μόνο η αλληλεγγύη και η συνεργασία, αλλά και σεβασμό προ τι αγορέ και σεβασμό προ τι οικονομικέ αρχέ, τι αρχέ οικονομία. Πρέπει να εντοπίσουμε τι ανάγκε βελτιστοποιώντα ε, τι δυνατότητε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να έχουμε το πιο αποτελεσματικό κόστος για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα αξιολογήσουμε φυσικά τις τροπολογίες ως προς αυτά που ανέφερα. Ευχαριστώ. Μισελ παρακαλώ. Έχετε τον λόγο ως και Μίχελ, Μίχελς ευχαριστώ. Η ε, κυρία Μίχελς, η ασφάλεια στην παροχή φυσικού αερίου και η διασυνοριακή αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Ιδιαίτερα τρεις παρατηρήσεις θα είχαμε. Η πρώτη, όσο και σημαντική να είναι η διασφάλιση φυσικού αερίου, αν έχουμε προβλήματα, η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να έχουμε τα ανανεώσιμα, ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, εγγενείς επιτόπιες ε, ενεργειακές πηγές και δυναμικό που πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει και αυτό να ενταχθεί στην πολιτική μας. Το δεύτερο και σε σχέση με τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν προηγούμενα και από τους σοσιαλδημοκράτες έχουμε κάποιες δυσκολίες με τα θέματα ορισμού κοινωνικών υπηρεσιών. Δεν έχουμε συμφωνήσει απόλυτα μεταξύ μας. Αν υποχρεωτικά αυτόν τον ορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα εγκρίνουμε ή μήπως θα ήταν καλύτερο να επαφεθεί το θέμα στα κράτη-μέλη. Μέχρι στιγμής αυτό θα προτιμούσαμε να γινόταν. Αν όμως από ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε κάτι και έχουμε και την τροπολογία 9 όπου γίνεται η απόπειρα να διαφοροποιηθούν κάποια πράγματα, αν το κάναμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρώ εγώ προσωπικά ότι το περιθώριο θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο. Κάνετε λόγο για θέματα ε, μέρημνας φροντίδας παιδιών και συναφή. Θα προτιμούσα Δηλαδή κάπως να εξειδικευθούν, να, είναι, να αποσαφινιστούν περισσότερο τέτοιου είδους προσεγγίσεις και θέματα. Το τρίτο, η τρίτη παρατήρηση είναι φυσικά η συμπερίληψη, η ένταξη των Δήμων και κοινοτήτων στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αν θέλουμε να περιφερειοποιήσουμε τις πολιτικές μας πρέπει στους εταίρους μας, οι εταίροι μας να είναι ε, σαφές ε, ποιες ε, προτεραιότητες, ποια δικαιώματα έχουν και ποια είναι η θέση τους. Συμφωνούμε όμως νομίζω σε μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις που εξετέθησαν. Thank uh, Σας ευχαριστούμε. Θα θέλατε να παρέμβετε εσείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριε ο Θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει απογοήτευση από πλευράς του συναδέλφου της ομάδας μας διότι δεν ήταν δυνατόν να προσέχει και να παρουσιάσει αυτά τα θέματα ο ίδιος. Είμαστε είναι γνώμων για το έργο και τις τροπολογίες Συμφωνούμε με το ότι το επίπεδο νομοθεσίας δεν διασφαλίζει τη σταθερότητα των αγορών φυσικού αερίου. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει εισαγωγή ενός νέου μηχανισμού, ενδυνάμωση των υφιστάμενων μηχανισμών ώστε να διασφαλιστεί ένα επαρκές επίπεδο προστασίας και για να ενθαρρυνθεί και η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Συμφωνούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργεί επαρκώς η αγορά ε, φυσικού αερίου και θα πρέπει γειτονικά κράτη να ε, προστατευτούν από πιθανώς αρνητικές επιπτώσεις. Πρέπει να διασφαλιστεί ανθεκτικότητα όσον αφορά περιπτώσεις διακοπής παροχής φυσικού αερίου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Λιθουανία που χρησιμοποιείται μόνο από κατά το 1 τρίτο του δυναμικού του αυτός ο σταθμός. Για διαφορετικούς λόγους βέβαια αυτό. Θα μπορούσαμε πολύ περισσότερο να κάνουμε χρήση αυτού του τερματικού. Και αντί να ομιλήσω διαζώσεις ε, σήμερα επ' αυτού, αυτό που χρειαζόμαστε είναι το North Stream 2 και το North Stream 1 που ε, χρησιμοποιείται μόνο κατά το ίμιση του δυναμικού του. Και γνωρίζουμε ότι τα ανανεώσιμα και η πράσινη ενέργεια όλο και περισσότερο απαιτείται να χρησιμοποιούνται και γι' αυτό η κατανάλωση φυσικού αερίου δεν θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, σε μεγαλύτερο βαθμό. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα θέμα που είναι θετικό για θέματα ενέργειας πολλοί πολίτε αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εξόφληση λογαριασμών φυσικού αερίου κατά το χειμώνα ιδιαίτερα λόγω υψηλών δαπανών, υψηλών ε, λογαριασμών ε, υφίστανται μεγάλα προβλήματα αυτές οι οικογένειες, αυτά τα νοικοκυριά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρξουν πρόσθετες ρήτρε ασφάλειας ώστε να αντιμετωπίσουμε, να αποφύγουμε την ενεργειακή φτώχεια εντό εισαγωγικών, την ενεργειακή παινία. Επιτρέψτε μου να στρέψω την προσοχή σας στο τεράστιο δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, σε σχέση με, την, <clears throat> με τα ορυκτά. Η χρήση ε, ορυκτών ε, για ενεργειακούς σκοπούς μπορεί να γίνεται για να προστατέψουμε την Ευρώπη, να προστατευτούμε από εξωτερικούς παρόχους ε, ενεργειακών προϊόντων. Όλα αυτά, μιλώντας για ενεργειακή αποδοτικότητα, πρέπει να αξιολογηθούν όχι σε σχέση με τη μείωση του κόστους ενέργειας. Ως πρώην δήμαρχος θα έπρεπε να πω ότι είναι δυνατόν να μειωθούν οι δαπάνες για θέρμανση νοικοκυριών. Εμείς ε, έχουμε μειώσει ε, κατά το ίμιση τις ε, δαπάνες αυτές και πρέπει να διασφαλιστούν όλοι οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις ώστε η χρήση να ανταποκρίνεται και να συνάδει με τους στόχους του ορίζοντα 2020 και να υπάρχει συνέργεια σε σχέση με άλλα μέσα. Πρέπει να ανανεωθεί και να ενδυναμωθεί η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών που είναι σχεδόν ανύπαρκτη σήμερα. Πρέπει να ευελτιωθούν οι υποδομές για τις μεταφορές και εξ του εισηγητή των Πρασίνων θα ήθελα να ευχαριστήσω και ελπίζω ότι θα εξευρεθούν οι αναγκαίοι συμβιβασμοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, βλέπω την κυρία Ντεμάτο. Ίσως θα μας παρουσιάσει την άποψή έτσι μετά. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μόζερ από την ε, ε, Γενική διάθεση Ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Πρόεδρε που με καλέσατε σήμερα το πρωί. Η ε, ενεργειακή ασφάλεια είναι ένας από τους πέντε πυλώνες ε, της Ενεργειακής Ένωσης που αναφέρεται βεβαίως ιδιαίτερος και στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές με περιλαμβανομένου και του βιοαερίου το οποίο αναφέρεται και στην ε, συζήτησή σας και συνδέει επομένως την τωρινή συζήτηση ε, με τη συζήτηση για τις ε, ανανεώσιμες πηγές η ενεργειακή ασφάλεια θα καλυφθεί αργότερα πάντως με άλλη απόφαση. Το φυσικό αέριο θα παίξει σημαντικό ε, ρόλο όποιο, και, όποιο σενάριο και αν επιλεγεί για την περίοδο 20-25. Και επομένως είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να πούμε ότι είναι το πιο καθαρό ε, ορυκτό καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια μιας οικονομίας μετάβασης προς χαμηλή χρήση <clears throat> άνθρακα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η εσωτερική αγορά δεν μπορεί πάντα να λύσει όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι τούτος ο κανονισμός είναι απαραίτητος έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, αντιμετωπίσουμε ε, κρίσεις ε, ενεργειακές σαν αυτές του 6, του 9, του 14. Η προσέγγιση έχει εστιαστεί πολύ μέχρι τώρα ε, στις ε, εθνικές λύσεις, οι οποίες δεν λαμβάνουν ικανοποιητικά ε, υπόψη είναι το, το γενικότερο προβληματισμό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν και να θεσμοθετηθούν διασυνοριακά μέτρα και ότι η ανάλυση πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνεται από κοινού. αυτή η ανάλυση δεν μπορεί να ε, σταθεί από μόνη της, δεν είναι ικανή και αρκετή και επομένως ε, χρειαζόμαστε ε, την δημιουργία ενός σωστού μηχανισμού. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τα θέματα αυτά που είναι τόσο σοβαρά σε ad hoc λύσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια, ένας σωστός ορισμός από τον Ευρωπαίο Νομοθέτη και από το ε, Συμβούλιο. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένα κριτήρια για τη σύσταση των περιφερειών Θέλουμε τα, οι ομάδες να είναι σταθερές ε, και ε, ε ολιγάριθμες, ε, να δημιουργηθούν επομένως συνέργειες οι οποίες θα χρησιμοποιούν τα ισχυρά σημεία και θα καλύπτουν τα ασθενή σημεία των κρατών και με τον τρόπο αυτό ε, να καλύπτονται τα προβλήματα όλων των χωρών. Οι ε, διάδρομοι επίγουσας ε, ανάγκης βεβαίως είναι καλό να υφίστανται αλλά δεν μπορούν να αποτελέσουν πανάκια και ε, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν αλλά αντιθέτως να ενισχύσουν τις περιφερειακές ε, ομάδες έτσι ώστε να διευκολύνουν το φυσικό αέριο το οποίο θα προωθηθεί από μια χώρα προς μια άλλη οποτεδήποτε μια τέτοια ανάγκη παρουσιαστεί. Η αλληλεγγύη είναι το δεύτερο πιο σημαντικό σημείο αυτού του ε, κανονισμού. Εδώ προβλέπεται ένας συγκεκριμένο μηχανισμός. Θα πρέπει να δούμε ποιες ε, ε, θα είναι οι ρυθμίσεις οικονομικές, διοικητικές ε, πρακτικές. Τον Σεπτέμβριο θα έχουμε ε, συνάντηση του συντονιστή, της συντονιστικής ομάδας με τα κράτη-μέλη και με τους εμπλεκόμενους. Ε, η ε, ευελιξία δεν είναι σημαντική βεβαίως, αλλά δεν μπορεί εξ αρχής να ρυθμίσει όλα τα στοιχεία. Ένα άλλο στοιχείο λοιπόν της δικιάς μας πρότασης είναι η διαφάνεια των συμβάσεων βάσει συγκεκριμένων ε, κριτηρίων. Γνωρίζουμε και μάθαμε από το, ε, τις παρελθούσες ε, ενεργειακές κρίσεις ότι τα κράτη-μέλη δεν είχαν πλήρη συνείδηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στις συμβάσεις τις οποίες υπέγραφαν και τις δυνατότητες υπέρβασης συγκεκριμένων ενεργειακών κρίσεων η βελτίωση της ε, ε, συνεργασίας ανάμεσα στην Ενεργειακή Επιτροπή ε, και τα συμβαλόμενα μέρη θα πρέπει να προωθηθεί έτσι και αυτό προς συμφέρον και των δύο πλευρών. Δεν θέλουμε ή δεν προβλέπουμε μία μονομερή βοήθεια προς την εσωτερική αγορά αλλά μία αμφίδρομη σχέση με την ενεργειακή κοινότητα. Uh, protected customers. Um, Οι προστατευόμενοι καταναλωτές, και ε, ε, ε υπηρεσίες ε, δημοσίου ενδιαφέροντος. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένος ορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, ε, ε, ένας ορισμός ο οποίος αφενός δεν θα δείχνει υπερβολική ανοιχτοχεριά, αλλά δεν θα δημιουργεί και προβλήματα στην σωστή λειτουργία των χωρών από την άλλη. Επίσης θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια στοιχεία καινούρια, όμως κυρίως θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ήδη υπάρχουσες δομές ενδεχομένως ε, ε, δημιουργώντας ε, κάποιους ευρύτερους διαδρόμους ή έναν ευρύτερο ορίζοντα. Ναι, είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε αμφίδρομες ροές σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο, κυρίως όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την δυνατότητα παροχής αερίου σε γειτονικές χώρες. Αυτά και σας ευχαριστώ. Κύριε Πορέμπα, θέλετε τον λόγο. Ε, να πω δύο λόγια για να ολοκληρώσω συνοψίζοντας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα σας τα σχόλια, όλες τις παρατηρήσεις σας και προτάσεις σας. Θεωρώ ότι οι προτάσεις σας θα εμπλουτίσουν και θα ενισχύσουν τη γνωμοδότησή μου ως τροπολογίες Υπάρχει λοιπόν αυτή η γενική συνένεση και ε, ότι χρειαζόμαστε πρόσθετα μέτρα για τη διεύρυνση αυτού του πλαισίου και διασφάλιση μιας καλύτερης παροχής φυσικού αερίου στην ε, κοινή αγορά. Και θεωρώ, και αυτό είναι ικανοποιητικό, και θεωρώ ότι τρεις θα πρέπει να είναι οι άξονες που θα μας βοηθήσουν να το πετύχουμε. Πρώτον, η περιφερειακή προσέγγιση. Δεύτερον, η έκφραση αλληλεγγύης. Και τρίτον, αλληλεγγύη φυσικά μεταξύ των ε, επιμέρους κρατών μελών. Και τρίτον, διαφάνεια συμβάσεων. Θα ήθελα λοιπόν να χρησιμοποιήσω αυτά τα τρία στοιχεία ως ε, βάση της γνωμοδότησής μου Είμαι ανοιχτός για τις τροπολογίες που θα μπορούσαν να κατατεθούν στα θέματα που αναφέρθηκαν, ευθυγραμμιζόμενοι βέβαια με τα θέματα τα οποία προαναφέραμε στην ε, παρουσίασή μας, δηλαδή τους τρεις κύριους άξονες που θα ήθελα να συμπεριληφθούν σε αυτή τη γνωμοδότησή μου. Θέλω για άλλη μια φορά σας ευχαριστήσω πολύ και για ε, επίσης να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι αυτή η γνωμοδότηση που από κοινού θα συντάξουμε θα είναι μια γνωμοδότηση που στο τέλος τέλος ε, θα προσφέρει στην Επιτροπή Περιφερικής Ανάπτυξης ε, ένα αίσθημα θετικό ότι συνεισφέρει και συνεισφέρει θετικά στη δημιουργία αυτών των σχέσεων που σίγουρα θα μας δώσουν τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε μια βελτιωμένη παροχή φυσικού αερίου για το σύνολο της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης μια παρουσίαση από το Τμήμα Πολιτικής Β για τις υπηρεσίες κοινή ωφέλεια κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020. Η Επιτροπή μας συζήτησε αυτή τη μελέτη για να δούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το, ε, ε, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά κονδύλια για τέτοιες επενδύσεις στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Η μελέτη είχε προετοιμαστεί και σήμερα θα δούμε τα αποτελέσματά της. Θα τα παρουσιάσει ο κύριος Ερικ Γκλέρσεν, ανώτερος σύμβουλος. Μετά την παρουσίαση θα δώσω τον λόγο στους βουλευτές ε, για ερωτήσεις και σχόλια. Τώρα κύριε Γκλέρσεν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές, κύριε και κύριοι, σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μα δίνετε να παρουσιάσουμε αυτή την μελέτη μας ε, για τις υπηρεσίε κοινή ωφέλεια. Το... Οι υπηρεσίες αυτές στο πλαίσιο τη συνοχή είναι και πρόκληση και παράδοξο. Είναι πρόκληση για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο ποσοστό της ε, πολιτικής ε, συνοχής άμεσα ή έμεσα συνδέεται με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Δεύτερον, σπάνια χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό στο πλαίσιο της ε, πολιτικής συνοχής. Είναι ο όρος της πολιτικής ανταγωνισμού και ακριβώς ε, στόχο έχει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ υπηρεσιών κοινή ωφέλεια και διατήρηση του ανταγωνισμού. Και εδώ πέρα ακριβώς βρίσκεται το παράδοξο, γιατί οι υπηρεσίες αυτές έχουν μεγάλη σημασία για την οικονομική και κοινωνική συνοχή και την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη και μπορεί η πολιτική συνοχή να συνεισφέρει σε αυτό, αλλά δεν αναφέρεται συχνά. Τι είναι λοιπόν οι υπηρεσίες κοινή ωφέλειας. Μιλάμε εδώ πέρα λοιπόν για τις υπηρεσίες ε, οικονομικής, οικονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή ε, έχουμε οικονομικές δραστηριότητες σε ένα πλαίσιο αγοράς ε, που έχουν αποτελέσματα προς ε, το γενικό συμφέρον που δεν θα ε, παρέχονταν χωρίς ε, κάποια δημόσια παρέμβαση. Υπάρχει βέβαια εδώ πέρα μια ταυτολογία. Οπότε η αιτιολόγηση του πεδίου παρέμβασης είναι πράγματι μια ταυτολογία. Μετά η έννοια του δημοσίου συμφέροντος δεν είναι ούτε κάτι το απλό ούτε κάτι το στατικό οι ανάγκες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, από κοινωνική ομάδα σε κοινωνική ομάδα και επίσης εξελίσσονται μες στον χρόνο. Όπως ε, μας έδειξε η συζήτηση για την ευρυζωνικότητα ή τα κινητά τηλέφωνα, αν πρέπει να θεωρηθούν υπηρεσίες κοινή ωφελής. Επιπλέον, το πλαίσιο της αγοράς ε, στο οποίο οι δημοσιοφορείς μπορούν ή δεν μπορούν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες εξελίσσεται ειδικά στο πλαίσιο της παγκόσμιας ρύθμισης ή απορρίθμισης οπότε πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυναμικό πεδίο και έτσι χρειάζονται συνεχώς ενημερώσεις. Στην σύντομη αυτή παρουσίαση θα εξετάσουμε πρώτα απ' όλα την παροχή υπηρεσιών κοινής μετά θα δούμε την συνεισφορά που κάνουν τα Ευρωπαϊκά Διαστρωτικά Ταμεία και τις συστάσεις μας. Πρώτα απ' όλα, τι είναι η υπηρεσία κοινή ωφέλεια στην Ευρώπη. Είναι μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι συνολικά 25% της προστεμενης αξίας, 30% της απασχόλησης, 22% όλων των επενδύσεων. Ε, αυτά βεβαίως διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όταν μιλάμε για προσθέμενη αξία, είναι λιγότερο από 20% στη Ρουμανία, αλλά πάνω από 30% σε Βέλγιο, Δανία, Πορτογαλία, Γαλλία. Οπότε εδώ διαφέρει η προσθέμενη αξία. Το ίδιο και η απασχόληση. Κάτω από 19% στη Ρουμανία, πάνω από 30% στη Σουηδία και Βέλγιο. Και όσον αφορά τις επενδύσεις πηγαίνουμε από 11% σε Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα 60% στην Λιθουανία. Βλέπουμε λοιπόν μεγάλες διαφορές. Επίσης παρατηρούμε την περίοδο 2006-2010 πως το, η σχετική τους σημασία εντός της οικονομίας αυξάνεται, οπότε παίζουν ένα σταθεροποιητικό ρόλο σε περιπτώσεις κρίσης. Χοντρικά λοιπόν παρατηρούμε πως η πολιτική αυτή αφορά το 1 τέταρτο της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι κάπως δύσκολο να μιλήσουμε για μια κατηγορία χάραξης πολιτικής όταν μιλάμε για κάτι τόσο μεγάλο. Ταυτόχρονα μπορεί κανείς να πει ότι ε, είναι ο κλάδος ε, χάραξης πολιτικής όπου καθορίζεται η ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της αγοράς. Όπως ξέρουμε η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ασχολείται με φορολογικά ζητήματα, δεν ασχολείται με ζητήματα μισθολογικά, το δικαίωμα της απαιτίας κτλ. Όμως λαμβάνει μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει την δυνατότητα στις τοπικές και εθνικές αρχές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών. Μιλάμε για τον ορισμό δηλαδή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Στην διαδικασία αυτή βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανισορροπία βλέπουμε πως ε, η δυνατότητα σύστασης κοινών ευρωπαϊκών λύσεων είναι κάτι το δύσκολο και δυσκίνητο ταυτόχρονα ή αποφάσεις για την ε, υπεράσπιση άνθρα ατομικών δικαιωμάτων ε, για κινητικότητα και εμπόριο τα οποία πιθανώς παραβιάζονται από τη συνθήκη λαμβάνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης βλέπουμε πως είναι ένα τόσο διαφοροποιημένο πεδίο, ώστε δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε κάποιες γενικέ αρχές. Υπάρχουν όμως δύο βασικοί τρόποι να δούμε τι υπηρεσίε κοινή ωφέλεια. Ο ένας είναι να ρυθμίσουμε την αγορά ευθύ εξ αρχή και να πούμε ότι πρέπει η αγορά να υπάρχει σε ένα πλαίσιο. Ο άλλο τρόπος είναι να δούμε τι αποτελέσματα έχει η λειτουργία τη αγορά και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα αρνητικά. Και αυτή είναι η βασική προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα με την εξαίρεση κάποιων κλάδων με μεγάλες δημόσιες επενδύσεις όπως η ενέργεια ή οι μεταφορές. Ποια είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή τα βασικά ζητήματα της παροχής τέτοιων υπηρεσιών στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, η βελτίωση των πρακτικών εξωτερικής ανάθεσης. Όπως ξέρουμε αυτό χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο Βλέπουμε πως ε, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί βεβαίως περιορίζουν εδώ πέρα τα πράγματα λόγω του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Το ασφαλέστερο που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αρχή είναι να αναζητήσει εξωτερική ανάθεση σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό για να αποφευθεί οποιαδήποτε υπόνοια κρατικής ενίσχυσης. Επίσης υπάρχουν προβλήματα με την εξωτερική ανάθεση, ειδικά για τοπικές και περιφερειακές αρχές και πάντα χρειάζεται ένα πλαίσιο για να γίνει αυτό. Στο πλαίσιο αυτό επίσης ε, σημαντικό είναι το θέμα της ποιότητας των υπηρεσιών. Υπάρχουν στοιχεία ποιότητας όπως ε, παραδείγματος χάρη το να είναι πρόσιτες οι τιμές ε, και δίκες, κατά οποίο συχνά βεβαίω οι ιδιωτικές εταιρείε δεν εξετάζουν. Ένα βασικό ζήτημα είναι πώς θα οικοδομηθούν ΣΔΙΤ που θα εκπληρώνουν όλες ε, τις προσδοκίες που υπάρχουν για την παροχή δημοσίων αγαθών. Ξέρουμε τώρα πως υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Κομισιόν ένα κέντρο εμπειρογνωμοσύνης ΣΔΙΤ. Η συμπερίληψή τους όμως πάντα ήταν προβληματική λόγω ρυθμιστικών περιορισμών. Τρίτον, έχουμε το ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κοινωνική επιχειρηματικότητα που παίζει μεγάλο ρόλο στην παροχή ε, υπηρεσιών κοινή ωφέλη, καθώ ειδικά στην περίοδο τη κρίση σε κάποιε χώρε αποδείχθηκε πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρχει ένα σταθερότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για να αναπτυχθεί. Τέταρτον, μια πρόκληση για πολλές τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι μια δημοκρατική πόλωση του πληθυσμού ή και συρρήκνωση, επειδή αυτό σημαίνει με διαφορετικές ταχύτητες και σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης η ανταλλαγή εμπειριών για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την συρρήκνωση για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και στη γύρανση και στην αλλαγή του πληθυσμού ε, είναι κάτι το σημαντικό. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανταλλαγής εμπειριών εδώ πέρα και το τελευταίο σημαντικό ζήτημα που θα ανέφερα είναι η διασυνοριακή παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Μπορεί να σημειωθεί μεγάλη πρόοδος ακόμα σε αυτό το μέτωπο και είναι πολύ βασικό για το ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή πώς θα ξεπεράσουν ρυθμιστικά, πολιτιστικά και γλωσσικά εμπόδια μεταξύ κρατών μελών. Αν δούμε τώρα τις ε, συνεισφορές ε, των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, κυρίως ε, αυτά ενισχύουν τις επενδύσεις, όχι την παροχή υπηρεσιών. Βλέπουμε επίσης πως υπάρχει η αρχή της συγκέντρωσης των προσπαθειών μέσω των θεματικών στόχων, οπότε περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής και παροχής τέτοιων υπηρεσιών. Π.χ. δεν βλέπουμε πώς θα μπορούσε η εκπαίδευση να βοηθήσει την αγορά εργασίας να λειτουργήσει. Μια τέτοια διαρθρωτική συνεισφορά των υπηρεσιών κοινή ωφελίας δύσκολα θα ενταχθεί στους θεματικούς στόχους του κάθε προγράμματος. Μετά βλέπουμε πως δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμιστικές προβλέψεις για έργα τα οποία σχετίζονται με υπηρεσίες κοινή ωφέλεια. Οπότε... Βλέποντας τις ιδιαιτερότητες του πώς λειτουργούν αυτά, πώς ε, εφαρμόζονται, αυτά δεν έχουν περιληφθεί στους σχετικούς κανονισμούς. Επίσης, βλέπουμε πώ είναι στους σχετικους κανονισμους επισης βλεπουμε πως ειναι σημαντικό ο ρόλο. Ε, των ε, διεθνών ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας που παίζουν ε, σημαντικό ρόλο στην αύξηση της γνώσης ε, των βέλτιστων πρακτικών. Όταν παρατηρούμε λοιπόν τις βέλτιστες πρακτικές υπάρχουν κάποια κέντρα που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν π.χ. Στην ε, Βόρεια Σουηδία υπάρχουν κάποια διεθνή κέντρα επανεκπαίδευσης ανθρώπων για να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά και μεταξύ τους Αργεμίν και της Ζάρλαντ στα γαλλογερμανικά σύνορα υπάρχει κοινή διαχείριση βιολογικού καθαρισμού που είναι αποτέλεσμα δεκαετιών συνεργασίας και υπάρχει η πρόκληση του να φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα μέσω προγραμμάτων, τα οποία όμως προγράμματα περιορίζονται σε λίγα χρόνια. Ενώ εδώ πέρα μιλάμε για βάθος δεκαετιών για παροχή υπηρεσιών κοινή ωφέλεια. Αυτή είναι η παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε με βάση τις βέλτιστες πρακτικές. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο πώς λειτουργούν οι συνεισφορές των διαρθρωτικών προγραμμάτων με βάση κάποια παραδείγματα. Βλέπουμε εδώ πέρα το πώς λειτουργεί ο κανονισμός ε, από τον κανονισμό στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, ας αναφερθούμε τώρα στις εργατικές κατοικίες στη Μάλτα. Υπάρχει μία προτεραιότητα η οποία λέγεται αναζωογόνηση ε, κοινοτήτων οι οποίες ε, ύστερούν και το νόημα εδώ πέρα ήταν στη Μάλτα να οικονομηθούν ποιοτικέ εργατικέ ε, κατοικίε. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα έλεγε ότι αυτό θα γινόταν μέσω ανακαίνηση δημοσίων χώρων ε, και των εργατικών αυτών κατοικιών ε, στο λιμάνι της Βαλέτας. Και η λογική ήταν ότι μέσω των επενδύσεων αυτών θα υπήρχαν θετικά αποτελέσματα στην υγεία και στην κοινωνική ένταξη. Αν ε, προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το σκεπτικό, βλέπουμε πως υπάρχει πάλι μια ταυτολογία που ανέφερα και στην αρχή. Δηλαδή, η παρέμβαση των ευρωπαϊκών κονδυλίων έχει σημασία όσο ε, στο μέτρο που παρεμένει στο κομμάτι εκείνο της ε, αγοράς στέγης που έχει αρνητική επίδραση στην κοινωνική ένταξη. Αν ο στόχος λοιπόν είναι η κοινωνική ένταξη και η υγεία, μπορούμε να αμφισβητήσουμε, να θέσουμε το ερώτημα πως ε, άλλες παρεμβάσεις θα ήταν πιο αποτελεσματικές αντί να εστιαστούμε σε μια συγκεκριμένη γειτονιά της κεντρικής ε, βαλέτας. Ίσως ε, η λογική ήταν να υπάρχει η μεγαλύτερη ανάμειξη εργατικών κατοικιών και μη. Και έχει κανείς την εντύπωση ότι το σκεπτικό της πολιτικής ανταγωνισμού επικρατεί στην πολιτική συνοχής. Δηλαδή έχουμε μια συγκεκριμένη λογική για την πολιτική ανταγωνισμού αλλά όχι για τις υπηρεσίες κοινή ωφέλεια. Π.χ. εδώ πέρα υπάρχει μια παρέμβαση στην αγορά στέγης και υπάρχει, γιατί υπάρχει μια αρνητική επίδραση της ελεύθερης αγοράς, δηλαδή ότι έχουμε υποβαθμισμένες κατοικίες. Αντί να πούμε πως έχουμε στόχους ε, εδαφικής ε, συνοχής που μετά θα όριζαν τη λογική της παρέμβασης. Επειδή αυτό δεν έχει γίνει λοιπόν, καταλήγουμε σε μια παρέμβαση η οποία είναι μια παρέμβαση σε μια γειτονιά που εντάξει μπορεί να είναι απόλυτο θεμητό να βελτιωθεί μια γειτονιά της ε, Βαλέτας, αλλά αυτό είναι συνεπές με την λογική που υπήρχε. Ένα άλλο παράδειγμα. Η ευρυζωνικότητα στην Εστονία. Υπάρχει μια προτεραιότητα επένδυσης, ε, π.χ. τα ευρυζωνικά δίκτυα, οδήγησε σε μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό έχει στόχο να βελτιώσει την κάλυψη ευρυζωνικότητας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για προώθηση της ψηφιακής οικονομίας και της ε, ανάπτυξης με βάση τη γνώση. Βεβαίω πάλι μπορούμε να πούμε πως η ευρυζωνικότητα θα δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείες να πάνε στην ψηφιακή οικονομία και να αναπτύξουν τη γνώση. Βεβαίως ε, βλέπουμε πως ε, καμιά φορά δεν είναι αυτός ο βέλτιστος τρόπος δημόσιας παρέμβασης. Δηλαδή το να προωθούμε τέτοιες δραστηριότητες θεωρούμε ότι οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση και άρα μπορεί μετά να ακολουθήσει η ιδιωτική πρωτοβουλία για να παρέχει ευρυζωνικότητα. Οπότε δεν είναι να εστιαζόμαστε μόνο στις υποδομές. Και η λογική αυτή των υποδομών ε, πάλι όπως είπα προκύπτει από αυτή την ε, προσέγγιση της πολιτικής ανταγωνισμού που έχει μπει και στην πολιτική συνοχής. Πάντα δηλαδή λέμε ότι όταν δεν υπάρχουν υποδομές πρέπει να κάνουμε κάτι. Οπότε, να δούμε κάποιες από τις ελλείψεις. Βλέπουμε λοιπόν πως πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο οι λογικές των υπηρεσιών κοινή ωφέλειας προς την περιφερειακή ανάπτυξη και μπορούμε βεβαίως να δούμε την διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα, πάρα πολλά μέτρα τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να φτάσουμε σε, ένα πιο, σε μια πιο συνεκτική περιφερειακή ανάπτυξη και περισσότερη ευημερία στο περιφερειακό επίπεδο. Οπότε η εστίαση αυτής της υποδομές ε, μπορεί ακριβώς να αντιμετωπιστεί μέσω των ε, επενδύσεων αυτών. Επίσης παρατηρούμε πως παρά τις ε, προσπάθειες, ειδικά στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η προσέγγιση είναι εδαφική, αλλά συχνά ακολουθούμε μια τομεακή πρακτική, δηλαδή οι συγκοινωνίες ε, θεωρούνται συγκοινωνίες. Δεν κοιτάμε δηλαδή τα θέματα της ε, κινητικότητας, της κοινωνικής κινητικότητας κτλ. Βλέπουμε επίσης πως τα προγράμματα κοινωνικής συνοχής θα μπορούσαν να προωθήσουν υπηρεσίες ε, κοινή ωφέλεια με την εξαίρεση βεβαίω των διεθνών προγραμμάτων. Κάτι το οποίο είναι μικρό κομμάτι των επενδύσεων. Τι προτείνουμε λοιπόν για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Είναι πρώτα απ' όλα μέτρα ενημέρωσης προς τις διαχειριστικές αρχές, τις επιτροπές παρακολούθησης για να μπορέσουμε ακριβώς να ενσωματώσουμε το σκεπτικό των υπηρεσιών κοινή ωφέλειας για το πώς μπορούν δηλαδή αυτά να βοηθήσουν τις περιφέρειες στους στόχους τους για την περιφερειακή ανάπτυξη. Μπορούμε επίσης να διαδίδουμε τις ε, βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ε, για να μπορέσουμε ακριβώ να τα προσαρμόσουμε αυτά στο, στις διάφορες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες ε, που υπάρχουν. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να ενθαρρύνουμε τη χρήση υφιστάμενων μέσων για ολοκληρωμένες επενδύσεις. Για να κινητοποιήσουμε ακριβώς ε, τέτοια μέτρα στο επίπεδο των κοινοτήτων για να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίε κοινή με τρόπο πιο αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο. Τώρα, πέρα από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο υπάρχουν και άλλες προοπτικές θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε το σκεπτικό, όπως σας είπα, της πολιτικής ανταγωνισμού. Να δούμε δηλαδή τα ευρωπαϊκά κονδύλια από τη σκοπιά του δημοσίου συμφέροντος και να τα κατατάξουμε ανακλάδο, π.χ. μεταφορές, υποδομές κτλ. ή αναγεωγραφική ζώνη και μέσω των υπηρεσιών κοινή ωφελία ε, όπου ήδη συνεισφέρουν. Πρέπει λοιπόν τα ευρωπαϊκά κονδύλια να τα δούμε ως συμπλήρωμα της πολιτικής ανταγωνισμού. Δεδομένη του ότι έχει μια δική του λογική και βασίζεται σε αυτά τα δύο σκέλη. Επίσης θα πρέπει να είναι λιγότερο τομεακή η προσέγγιση στην πολιτική ανταγωνισμού και θα πρέπει να παρακολουθούμε την παροχή υπηρεσιών κοινή ωφέλεια στο επίπεδο κάτω από αυτό της περιφέρειας ε, γιατί οι περιφέρεια είτε σε ΝΑΤΣ 3 είτε σε ΝΑΤΣ 2 κρύβουν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ δήμων, γειτονιών και η αύξηση της παρακολούθησης ε, θα καθιστούσε πολλά ζητήματα πιο ε, ορατά και επίσης ε, θα μας έδειχνε γιατί κάποιες περιφέρειες δεν μπορούν να φτάσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα ανάπτυξης. Μετά υπάρχουν πολλές δυνατότητες πρόληψης παροχής ε, διασυνοριακών τέτοιων ε, υπηρεσιών. Μπορούμε επίσης να συνεχίσουμε την οργάνωση βέλθων πρακτικών στο πεδίο των υπηρεσιών κοινή ε, ωφέλειας, να ενθαρρύνουμε τον διάλογο μεταξύ των ε, κύριων ε, διαρθρωτικών προγραμμάτων και των υπηρεσιών κοινή ωφέλης. Ήδη βλέπουμε στο πλαίσιο των μακροπεριφερειακών στρατηγικών κάποια σοβαρά πράγματα. Και βεβαίως υπάρχει ένα πλαίσιο διαλόγου για τις υπηρεσίες κοινή ωφέλειας. Π.χ. τα απόβλητα στην περιοχή Αδριατικής Ιωνίου. Ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ πέρα. Μετά, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας παροχής υπηρεσίας κοινή ωφέλεια σε ε, απομακρυσμένες περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού που κοστίζουν περισσότερο και είναι δύσκολο να δικαιολογηθούν σε καιρούς λιτότητας. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό σε σχέση με την προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το τι παράγουν αυτοί οι τόποι, σε σχέση με το κόστος. Και το να γίνει δηλαδή αυτή η αξιολόγηση του επιπλέον κόστους των υπηρεσιών κοινής οφειλίας σε σχέση με την προστιθέμενη αξία της παραγωγής μετά που ε, καθιστούν δυνατή. Και τέλος, πρέπει να δούμε το πώς ε, θα μπορούσαν τα διαρθρωτικά ταμεία να στηρίξουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Να έχει δηλαδή ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο να ληφθεί υπόψη. Να δημιουργηθούν ακριβώς αυτές οι ελάχιστες επενδύσεις για να ξεκινήσουν δραστηριότητε που βασίζονται σε εθελοντικές οργανώσεις και μη κερδοσκοπικές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία παρουσίασή σας, περιεκτική, γεμάτη στοιχεία πληροφοριακά. Κυρίες και κύριοι, τώρα μπορείτε να παρέμβετε. Θέλει κάποιος να παρέμβει. Νίλσον παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σου ειδικά και ούτως ή άλλως είναι κατανοητή η γλώσσα μου σε σχέση με το παρεμβαίνω. Δεν ήμουν στην Επιτροπή σε σχέση με την παρουσίαση της μελέτης, όμως θέλω να ευχαριστήσω. Διάβασα την περίληψη και είδα τα στοιχεία και ουσιαστικά η πείρα μου ως δημάρχου σε αυτό το κείμενο επιβεβαιώνεται με τα όσα διαπιστώνονται και για την οδό που θα ακολουθήσουμε σε σχέση με τα στοιχεία και τα προβλήματα που αναφέρονται στην έκθεση και μετά διατυπώνονται και κάποιες συστάσεις, θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και να πούμε ότι ίσως η πιο σημαντική, το πιο σημαντικό συμπέρασμα είναι ε, ότι ε, πρέπει κάποια σημεία να τα συμπτύξουμε και να τα ανακεφαλαιώσουμε. Καθίσταται με άλλα λόγια όλο και σαφέστερο ότι οι αρχές, οι δήμοι, οι κοινότητες όλο και περισσότερο εμπλέκονται στον ιδιωτικό τομέα και το έργο του, στο έργο του ιδιωτικού τομέα ευρύτερα. Και γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη αποδοχή και μεγαλύτερη συνοχή και συνεκτικότητα θα έπρεπε να δώσουμε κίνητρα για να γίνει κάτι τέτοιο σε μεγαλύτερο βαθμό. Είναι στο τέλος τέλος οι βασικές αρχές στις οποίες θεμελιώνεται η διαθωτική μας πολιτική και έχει θετική απήχηση αυτό. Και το λέγω και ως πρόεδρος της διακομματικής ομάδας για, αυτή, για αυτές τις πτυχές μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικότερο ρόλο αυτή η προσέγγιση σήμερα, πολύ σημαντικότερο από ό,τι μέχρι σήμερα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Χρειαζόμαστε όλο και λιγότερο τομεακά πιο εξειδικευμένες πολιτικές. Πρέπει πιο επικεντρωμένα να επικεντρωνόμαστε στην πολιτική συνοχής. Και αν το καταφέρουμε αυτό, καλύτερα συστήματα θα μπορούμε να οικοδομήσουμε, αποτελεσματικά προγράμματα και σχέδια που θα προαχθούν και που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα. Εμείς ως Επιτροπή Περιφερικής Ανάπτυξης θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουμε το ρόλο μας αυτό και να αφοσιωθούμε σε αυτό το έργο να σημειώσει πολύ προσεκτικά η γραμματεία αυτά και να προχωρήσουμε έτσι και στο τέλος τέλος να συνεργαστούμε και με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, την ΕΚΟΝ, την Οικονομική Νομισματική Επιτροπή και όταν έρχεται η ώρα να αξιολογήσουμε τα πράγματα θα μπορούμε πάντα να επισημάνουμε αυτή την έκθεση. Αυτή η έκθεση θα είναι πολύ χρήσιμη και σας ευχαριστούμε για Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος Μπόκοβιτς παρακαλώ. Σας, σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να πω, Πρόεδρε, ότι αυτή η μελέτη είναι πολύ σημαντική για το μελλοντικό μας έργο και τις μελλοντικές κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουμε στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής όπου πρέπει να προβληματιστούμε σχετικά με το μέλλον αυτής της ε, πολιτικής συνοχής. Συμφωνώ με εκείνους που λένε ότι η κοινωνική συνοχή πρέπει στην Ευρώπη να θεωρηθεί ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές υποθέσεις για το μέλλον μας, για το μέλλον της Ευρώπης. Και γι' αυτό είναι σημαντικό η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική και πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η κοινωνική συνοχή να διασφαλίζεται. Υπάρχουν παρόλα αυτά διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και υπάρχουν και μεγάλες διαφορές και στα ίδια τα κράτη-μέλη μας μεταξύ διαφορετικών περιφερειών. Από πλευράς μου με την πείρα δημαρχίας που είχα πρέπει να δούμε θεωρώ και την ποιότητα του δημόσιου τομέα και των δράσεών μας. Συχνά τόνισα ότι η ποιότητα του ε, δημόσιου τομέα πρέπει να αναβαθμιστεί και ότι έτσι θα μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε και τη φτώχεια. Και αυτό το δείχνει ανάγλυφα πολύ καλά και αυτή η έκθεση. Θα ήθελα να τονίσω τούτο. Το ότι δηλαδή η δημογραφική αλλαγή, οι δημογραφικές εξελίξεις ε, σε σχέση με τη δημογραφική μας δομή, οι προγνώσεις δεν είναι βίωνες. Ένα από τα κύρια συμπεράσματα είναι η υπεργύρανση του πληθυσμού της Ευρώπης. Υπάρχουν πολλά νέα μέσα τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πρέπει να τα εξεύρει και να τα χρησιμοποιήσει η Ευρώπη ώστε να δώσει μια απάντηση στα προβλήματα των δημογραφικών αλλαγών. Και η πείρα μας από τη Σλοβενία δείχνει ότι ε, οι οίκοι ευγυρίας στους οποίους ζουν ε, οι περίλικες οι οποίοι δεν μπορούν πλέον ε, να φροντίσουν τον εαυτό τους Παράλληλα όμως με όλα αυτά υπάρχει και η κατοίκον ε, ε, σύνδρομη, η κατοίκον βοήθεια. Μπορούμε έτσι να μειώσουμε σε τεράστιο ποσοστό το κόστος, διότι οι άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να στοχεύουμε και να εξοικονομούμε κονδύλια. Υπάρχουν πολλά τέτοια κέντρα και με τη δυνατότητα μείωσης του κόστους είχαμε θετικά αποτελέσματα. Οι άνθρωποι αυτοί απολαμβάνουν ενός αναβαθμισμένου επίπεδου ε, ζωής και διαβίωσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σπουδαιότητα οι κοινωνικές μεταφορές και μεταθέσεις και για τους ανέργους να επιτυγχάνονται προς κοινό όφελος. Και γι' αυτό στη Σλοβενία νέοι άνθρωποι, νέοι σκέπτονται πολύ συχνά, προβληματίζονται αν αξίζει τον κόπο να δουλέψουν και πολλοί από αυτούς αποφασίζουν να μην εργαστούν διότι θα έχουν κοινωνική υποστήριξη για τα παιδιά τους και οι κοινωνικές αυτές μεταφορές, μεταφορές κονδυλίων θα είναι προς όφελός τους υψηλότερες αν εργαζόντουσαν και έπαιρναν έναν σε εισαγωγικά χαμηλότερο μισθό. Θα έλεγα ότι εδώ ο, ο κρατικός τομέας, ο δημόσιος τομέας πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το κόστος, τα κόστη να μπορέσουν να μειωθούν Υποστηρίζω τέτοιου είδους μελέτες λοιπόν. Θεωρώ ότι οι βέλτιστες πρακτικές πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ μας ε, και σε σχέση με τις ε, συγκρίσεις ε, να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει συλλήβδη μία και μόνη μαγική λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πανενωσιακά θα έπρεπε να ισχύει, θα μπορούσε να λειτουργήσει θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών μας. Είναι καλή μελέτη και θετικό, θετική βάση για την... Ευχαριστώ. Κύριε Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω αγαπητέ κύριε για αυτήν την ε, ε, για αυτή την εργασία και πολύ σύντομα να πω την άποψή μου. Είναι περίπλοκες, οι όροι που έχουμε και οι προϋποθέσεις. Είναι περίπλοκοι, δεν λειτουργούν καλά και για να διορθώσουμε αυτά που δεν λειτουργούν δημιουργούμε νέους κανόνες που ενδεχομένως με τη σειρά τους ε, θα ε, δημιουργήσουν νέα προβλήματα. Πρέπει με πολύ απλό τρόπο να καθορίσουμε κάποιους όρους. Ευχαριστώ πολύ. είστε όντως πολύ σύντομοι. Ο κύριος Βανίστεν Ρόι. Ευχαριστώ. Στη σελίδα 118 και 119 βλέπουμε πράγματι την συγκεκριμένη σύνδεση μεταξύ των όσων ορίσαμε στον κανονισμό και των κομματιών εκείνων που αφορούν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Και αυτό είναι θετικό. Και βλέπουμε πως ε, και το Συμβούλιο στο 533 λέει πως οι κανονισμοί ακόμα δεν έχουν φτάσει ε, σε αυτή την σύνδεση της πολιτικής. Όπως είπε και ο συνάδελφος, ε, πρέπει και το ερώτημα απευθύνεται και στην δικιά μας την γραμματεία της Επιτροπής μας. όταν θα φτάσει η στιγμή της επικαιροποίησης θα πρέπει να δούμε τη λογική γιατί η πολιτική της συνοχής βεβαίως αφορά άλλε ε, επιτροπές αλλά υπάρχει κάποια στιγμή εντός της ε, τρέχουσας πραγματικής περίοδου για να το εντάξουμε αυτό γιατί για μένα δεν είναι τόσο ε, σαφές ε, το πώς θα γίνει αυτή η βαθιά αναθεώρηση της προσέγγισής μας και γνωρίζω βεβαίως πως ε, έχουμε διάφορους ε, κλάδους, την καινοτομία, την ενέργεια, όπου γίνεται λόγος από την Κομισιόν για τις κρατικές ενισχύσεις και τα πράγματα είναι πολύ ε, ακριβώς ε, καθορισμένα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πρέπει να δούμε το σύστημα ή να δούμε την καλύτερη παρακολούθηση και στήριξη αυτών που είπε παραδείγματος χάρη ο κ. Ε, Μπόγκοβιτς για διασυνοριακά ζητήματα και τέτοια πράγματα. Για να δούμε ακριβώς ε, ποια είναι η συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί σε αυτή την έκθεση. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα. Επίσης, ε, μιλήσατε για τις εργατικές ε, κατοικίες ε, που είναι πράγματι υπηρεσίε κοινή ε, ωφέλεια. Αλλά αν δούμε τι γίνεται σε κάθε χώρα, ε, το καθήκον αυτό ανατίθεται στον ιδιωτικό τομέα ή σε ημικρατικό τομέα ή αλλού είναι 100% στα χέρια του κράτους. Οπότε θα πρέπει ακριβώ να το δούμε για να μπορέσουμε να, να απαντήσουμε στο επίπεδο των κανονισμών. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω πως ε, ε, θα υπάρχουν προβλήματα. Θυμάμαι ακόμα την οδηγία Μπόλκενστάιν και δεν ξέρω αν μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε ε, η δοκιμή βεβαίως ε, για το εάν κάτι συμφωνεί με το δίκαιο του ανταγωνισμού θα πρέπει να υπάρχει, αλλά να μην είναι τόσο σοβαρή η εξάντερεσιμότητα, ώστε να μην απομείνει καμία δυναμική. Εν ολίγης, what's the next step. Και βλέπω και του συναδέλφου εδώ πέρα που χαμογελάνε. Έχουμε ήδη ένα πολύ περίπλοκο σύστημα που πρέπει να απλοποιηθεί. Να δούμε τι, πώς θα το κάνουμε αυτό, αγαπητοί συναδέλφοι. Σας ευχαριστούμε. Πολύ καλό. Ναι, Ροντρίγκες παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτή και να συγχαρώ επίσης, γιατί είναι μια από τις λίγες φορές όπου βλέπω σε, τέτοια, σε τέτοιες εκθέσεις να παρουσιάζονται υπερπεριφερειακές, υπεραπομακρυσμένες περιοχές. Και αυτές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, οι υπερπεριφερειακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφερειακή μας πολιτική. Υπό αυτό το πνεύμα λοιπόν μπορούμε, όπως καθορίζεται και από την συνθήκη στο άρθρο 349, να δράσουμε και θα ήθελα δύο ερωτήσεις να κάνω. Σε σχέση με τη σελίδα 139 υπάρχει μια παράγραφος που αφιερώνεται σε αυτές ε, τις περιοχές. Δύο ερωτήσεις άμεσες θέλω να διατυπώσω για περισσότερες αποσαφηνήσεις ε, είναι παράγραφοι και είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τι βρίσκεται πίσω από αυτές για μένα να μου δώσετε επεξηγήσεις πώς από πλευράς ευρωπαϊκής δράσης μπορεί να προκληθεί να δημιουργηθούν επενδύσεις ε, σε αυτές τις περιοχές διότι το κόστος είναι πολύ υψηλό σε αυτές τις περιοχές. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο του υπερβολικού, υπερβολικά υψηλού κόστους. Θα ήθελα να ζητήσω περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Γιατί δεν φτάνει μία παράγραφος να κατανοήσει κανείς το πρόβλημα αντιμετώπισης αυτών των επενδύσεων. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γκλώρασεν. Είστε έτοιμος να απαντήσετε στις ερωτήσεις οι οποίες υπευλήθησαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές ε, τις ερωτήσεις οι οποίες δείχνουν ότι παίρνετε σοβαρά υπόψη την ε, έρευνά μου. Ας πούμε, παράδειγμα των ε, ε, Κατο χωρών. Ε, υπήρχε ε, ήδη στην χώρα αυτή ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης. Η Κομισιόν δεν συμφωνούσε με αυτό και το γεγονός ότι προσαρμόστηκε λοιπόν ολόκληρο το σύστημα δείχνει ότι υπήρχε η διάθεση προσαρμογής προς τις ευρωπαϊκές προσταγές. Τώρα όσον αφορά την, ε, ε, την χωρική και ε, κοινωνική συνοχή, όντως αυτά είναι στοιχεία τα οποία οπωσδήποτε θα συνοδεύσουν και συνόδευσαν στην Ολλανδική περίπτωση αλλά και στην Σουηδική αυτήν την απορρίθμιση η πολιτική συνοχή και η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να ειδωθούν σαν δύο σκέλη επί των οποίων θα πρέπει να βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ να συμφωνήσω απολύτως με την ιδέα ότι εδώ ο κύριος εχθρός μας είναι ο χρόνος, δηλαδή ο, ε, ε, η ταχύτητα της, ε, αυτού του αποσυντονισμού μπορεί να είναι πολύ μεγάλος και το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον μπορεί κάποιος να ε, παραμείνει σωστός ακολουθώντας αυτόν τον ταχύ ρυθμό ε, απορρίθμισης. Το timing λοιπόν ε, και η εξισορρόπηση μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων είναι κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά τις πιο απομακρυμένες ε, περιοχές και τη σχετική ε, ε, διάταξη που αφορά τις περιφέρειες αυτές σε σχέση με τις υπηρεσίες κοινή ωφέλειας. Ναι, εκεί χρειάζονται μαζικές επενδύσεις όσον αφορά τώρα τις πρόνοιες δεν υπάρχει μια ε, γενική τέτοια διάταξη, αλλά παρόλα αυτά μπορεί ε, να ε, υπάρξει η εφαρμογή βελτίστων πρακτικών, έτσι όπως έχουν εφαρμοστεί ανάμεσα σε νησιά, ας πούμε, που έχουν λίγο πληθυσμό ή βρίσκονται πολύ μακριά κτλ. Ναι, μπορεί να υπάρξει διάλογος. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η λύση. Διάλογος, ανταλλαγή ε, ευρωπαϊκά πρότυπα ε, όσον αφορά μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, οι λύσεις οι οποίες έχουν προταθεί. Λέμε ότι όλοι θα πρέπει να έχουν ε, ίδια πρόσβαση, αλλά αυτό, πρόσβαση, αλλά αυτό ε, ε, πραγματικά δεν μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή, αν ζει κανεί σε ένα απομακρυσμένο μέρος ή σε ένα νησί, δεν μπορεί να έχει την ίδια ακριβώ πρόσβαση σε νοσοκομεία ή σε κάτι άλλο. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να, και στις περιοχές αυτές να διευκολυνθεί η διαβίωση μέσα από πρόσβαση ε, σε συνοχή, σε κοινωνικέ υπηρεσίε. Είναι αλήθεια ότι ένα ενιαίο μοντέλο δεν μπορεί να ισχύει για όλου. Ευχαριστώ. Οπωσδήποτε λέει η Πρόεδρος δεν ε, τελειώνει εδώ η συζήτηση. Η Κομισιόν να πάρει το λόγο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά δύο, δύο πόδια είπαμε και ένα σώμα. Τι θα γίνει όμως, ε, το κεφάλι δεν θα πάρει και το... Εγώ αυτό που θέλω είναι πολιτική συνοχή ε, η οποία να είναι καλύτερη, να οργανώνεται καλύτερα και να παραδίδεται στους πολίτες καλύτερα. Και επομένως η Κομισιόν δεν πρέπει να έχει το λόγο. Ωραία, θα δώσουμε τη δυνατότητα στην Κομισιόν να δει την έρευνα αυτή. Και άντε, ας της δώσουμε και το λόγο. Κομισιόν. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι μεγάλο και οπωσδήποτε χρειάζεται λεπτομερέστερη συζήτηση. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο κ. Φανίστερο όσον αφορά την περιπλοκότητα του, στοιχεί, του ζητήματος και, το, και όσον αφορά τα επιπλέον στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ε, προσθεθούν στα πλαίσια βέβαια της απλούστευσης που όλοι επιζητούμε. Ένα θέμα θέλω να αναφέρω. Ε, δυστυχώς ε, δεν ε, παρακολούθησα από την αρχή τη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα ε, σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει να παραφορτώσουμε την πολιτική συνοχή. Η οικονομική ε, ε, κοινωνική και εδαφική συνοχή είναι ε, μοιρασμένη αρμοδιότητα, είναι κοινή αρμοδιότητα και επομένως θα πρέπει να γίνει ένα συνδυασμός ανάμεσα στο τι κάνει η Ευρώπη και τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα αυτή η τριπλή συνοχή και είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Ας πούμε όσον αφορά τη στέγαση, εδώ έχουμε ένα τομέα αποκλειστικής των κρατών μελών. Αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει ευρύτερη συζήτηση πάνω στα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ λέει η πρόεδρο. Οπωσδήποτε αυτή δεν θα είναι η τελευταία ε, φορά και η τελευταία συζήτηση ε, που θα αναφερθούμε στην ε, μελέτη αυτή. Σας ευχαριστούμε. Προχωρούμε λοιπόν. Επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως αφορά το διορθωτικό στον κανονισμό 1303-2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κλπ. Πρόκειται για ένα διορθωτικό, <laughs> συγγνώμη, διορθωτικό ε, για λόγους γλωσσικούς και Την 6η Ιουνίου το λάβατε αυτό το διορθωτικό του έτους 2016. Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται 13 ε, τεχνικές ε, και γλωσσικές ε, διορθώσεις επί του κειμένου που είχε εγκριθεί το 2013. Πρόκειται ένα κείμενο το οποίο είχε ελεγχθεί από τις νομικές υπηρεσίες των τριών οργάνων. Η Γραμματεία του Συμβουλίου μας ενημέρωσε ότι ήδη τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει με το διορθωτικό Εμείς επίσης αποφασίσαμε στις 24-25 Μαΐου για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζαμε το διορθωτικό αυτό. Για μία ημέρα ακόμα έχετε προθεσμία να αντιδράσετε για το διορθωτικό αυτό. 12 το μεσημέρι αύριο ημέρα Παρασκευή 17 Ιουνίου λίγη η προθεσμία υποβολής ετοιμάτων. Ε, ελήψη τέτοιων ε, προτάσεων το διορθωτικό θα θεωρηθεί ε, αποδεκτό και θα ψηφιστεί τον Ιούλιο. Κύριε Μπέρκοβιτς, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλά να πω ότι το διορθωτικό αυτό ε, είναι απόρρια ε, ε, μακροτά της διαδικασίας και το, η Κομισιόν θα επιθυμούσε γρήγορη έγκρισή του πλέον γιατί διαφορετικά θα έρθει σε αντιπαράθεση ή θα δυσκολέψει άλλα νομοθετήματα. Θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν να το μελετήσετε προσεκτικά μεν αλλά να προχωρήσετε και γρήγορα δε. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έχουμε λοιπόν 24 ώρες μπροστά μας για να υποβάλουμε σχόλια και μετά θα ξέρουμε λοιπόν αύριο το μεσημέρι ποια είναι η θέση των μελών. Προχωρούμε λοιπόν, είμαστε στα διάφορα. Υπό τα διάφορα θέλετε να ε, ε, υποβάλλετε κάτι. Όχι. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι η προσεχή συνεδρίασή μας ε, θα λάβει χώρα τη 13η Ιουλίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι και ξανά από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 6.30 και θα συνεχιστεί την 14η Ιουλίου 2016 μόνο το πρωί από τις 9 μέχρι τις 12.30. Κλείνω λοιπόν ε, αυτήν την ε, ε, συνεδρίασή μας και παρακαλώ τους συντονιστές να παραμείνουν διότι θα συνεχίσουμε με την συνεδρίαση των συντονιστών αλλά και κλεισμένων των θυρών.